Dear Συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε. Έχουμε απαρτία. Να ξεκινήσω με ορισμένες ανακοινώσεις του Προέδρου όσον αφορά τις ε, αποφάσεις των συντονιστών που ελήφθησαν χθες. Σημείο 1. Ορισμός εισηγητών. Ο κύριος Χρυσόγονος οριστήκε εισηγητή για την υπεράσπιση της αστυλίας του κυρίου Μποργέζιο, η κυρία Φεράρα ορίστηκε εισηγήτρια για την άρση της αστυλίας του Τσάμπα Μόλναρ. Ο κύριος Σοβάσκι ορίστηκε εισηγητής για την, για την άρση της αστυλίας του Ρολάντα Πάξας. Η κυρία Ρέγνερ ορίστηκε εισηγήτρια για την αποκάλυψη πληροφοριών φόρου εισοδήματος για ορισμένες επιχειρήσεις και κλάδους και υποκαταστήματα. Δεύτερον, τα ψηφίσματα που, που προτάθηκαν με βάση το άρθρο 133 του κανονισμού σχετικά με την προστασία της εμπιστευτικότητας των δημοσιογραφικών πηγών από τον Dominic Bild και αποφασίστηκε να προσκληθούν οι συντάκτες της ε, ε, έκθεσης. Της έκθεσης στο Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα σε σχέση με το, δικαίωμα, με το δίκαιο των επιχειρήσεων, με το Δικηγορικό Σύλλογο Παρισίων, ε, την Ένωση Δικηγορικών Συλλόγων της Γαλλίας κτλ. σε μελλοντική συνεδρίαση. Και τέταρτον, συμφωνήθηκε να αναβληθεί η πρόσκληση της, προς την Κομισιόν σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση για την αποκάλυψη ορισμένων πληροφοριών μη οικονομικής ε, φύσης από ορισμένες ε, μεγάλες επιχειρήσεις έως την συνεδρίαση της Επιτροπής 13 και 14 ε, ε, Ιουνίου. Επίσης, ε, για τη δικαστική εκπαίδευση με διασυνοριακές επιπτώσεις. Ο κύριος ε, ε, Ράντιεφ είχε προτείνει αυτό το θέμα από το ΕΛΚ, εγκρίθηκε και εγκρίθηκαν και κάποιες δράσεις που προτάθηκαν από τους σοσιαλιστές σχετικά με τις εταιρείες θηρίδας και με βάση πρόταση των Πρασίνων ελήφθη μια απόφαση για ένα σχετικό θέμα. Ε, επίσης, ε, θα συζητηθεί στην Επιτροπή μας το θέμα της βιοτεχνολογίας και της αντίστοιχης οδηγίας και θα προσκληθεί η Επιτροπή Άγκρη. Τέλος, θα συζητηθεί η Διοργανική Συμφωνία για την Καλύτερη Νομοθεσία. Η κυρία Κάουφμαν από τους Σοσιαλιστές η κυρία Ντίστρομ για το ΕΛΤΕ, η κυρία Χάουταλα από τους Πράσινους, ο κύριος Χρυσόγονος από την ΚΟΕ και ο κύριος Μποτόσκε από το ECR θα συμμετέχουν στη σχετική ομάδα εργασίας. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις του Προέδρου. Δεν βλέπω να υπάρχουν σχόλια, οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε με την μερίσια διάταξή μας με τα σημεία 17 και 18. Εγώ είμαι εισηγητής και θα μιλήσω τσεχικά. Ε, λοιπόν, εδώ έχουμε να κάνουμε με μία πρόθεση μια έκθεση σχετική με την κύρωση από τα κράτη-μέλη προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Διεθνούς Συμβάσεως για την ευθύνη και αποζημιώσεις για ζημία σχετιζόμενη με τη θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών με εξαίρεση της πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις. και επίσης σε δεύτερο στάδιο με τις πτυχές της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις. Προθεσμία για την κατάσταση των τροπολογιών 27 Μαΐου. Πρόκειται για μεσοπρόθεσμη, όπως είπα, έκθεση. Με στόχο να προβλεφθούν οι θέσεις του Συμβουλίου και της Κομισιόν, να ζητηθεί δηλαδή η ανάληψη πρωτοβουλειών για τροποποίησης. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την οδηγία που αφορά το περιβάλλον και διεθνείς συμβάσεις. Η διάμεση έκθεση στόχο έχει να καταγράψει τα αρνητικά στοιχεία που απορρέουν από τα κείμενα αυτά να προσδιορίσει την νομική βάση και τα διάφορα συστήματα ευθύνης σε περίπτωση ζημίας κατά τη μεταφορά από θαλάσσιες επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών. Αυτή είναι η ουσία και ξαναμετατρέπομαι σε πρόεδρο για να δώσω το λόγο στους συναδέλφους αλλά και την Επιτροπή, γιατί ίσως κυρία Τσαρούχα θέλει να λάβει το λόγο. Good morning. Thank you. Καλημέρα σας και ευχαριστώ. Η Επιτροπή καλωσορίζει την έκθεση, το σχέδιου εκθέσεως και ιδιαίτερα όσον αφορά τις ανησυχίες που έχει και η Επιτροπή εκφράσει σε αλλά και ο κλάδος ε, στην επιστολή, στην υποσημείωση παριθμών 1 στο σχέδιο της ενδιάμεσης έκθεσης του εισηγητή, δηλαδή επιφυλάξει σε σχέση με την νομική βάση για τις ε, πτυχές που δεν έχουν να κάνουν με τις αστικές υποθέσεις, δικαστική συνεργασία σε μη αστικές υποθέσεις. Και επίσης όσον αφορά την υποχρέωση κύρωσης από τα κράτη-μέλη του πρωτοκόλλου. Η Επιτροπή εν γέννη, όπως ε, σημείωσε και ο εισηγητής υπογραμμίζει την ανάγκη να είναι ομοιόμορφο, ενιαίο και όχι κατακαιρματισμένο το ευρωπαϊκό δίκαιο και για τους κανόνες που διέπουν τα δικαιώματα των θυμάτων ε, ρηπάνσεως και τις υποχρεώσεις των φορέων ε, της βιομηχανίας. Βεβαίως είμαστε διατεθειμένοι να προχωρήσουμε στη συνεργασία με το Συμβούλιο σε περαιτέρω εξέταση και των εγγράφων και σε διευκρίνηση, αν μου επιτρέπετε, για την παράγραφο H ήταν του σχεδίου μου σε προθέσμους εκθέσεως της 135 την πρόταση δηλαδή για πτυχές δικαστικής συνεργασίας εκτός αστικών υποθέσεων Η ELD αποκλεί από το πεδίο εφαρμογή τη ε, περιστατικά που θα υπάγονταν στη σύμβαση AHS. Ε, Και αυτό μόνο περιστασιακά. Αυτό δηλαδή δεν σημαίνει ότι αν ε, κυρώσει το πρωτόκολλο ένα κράτος μέλος δεν θα εφαρμόζεται η ELD στο εν λόγω κράτος. Σε περίπτωση περιστατικού δηλαδή που προκύπτει ρήπανση τα εθνικά δικαστήρια μπορούν να προσδιορίσουν ότι το περιστατικό έχει ε, λόγο να υπαχθεί στο, στη Σύμβαση HNS υπό το πρωτόκολλο του 2011 και άρα ισχύει η νομοθεσία όπως Αυτή είναι η αδικοπρακτική ευθύνη, μάλλον είναι η αστική ευθύνη χωρίς αδικοπραξία. Εν προκειμένου, όπως συμβαίνει άλλωστε και με τις άλλες ε, συμβάσεις του πρωτοκόλου της σχετικής με τη θαλάσσια ρήπανση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Άντερσον. Ευχαριστώ. Καλή έκθεση. Λέει τα σωστά πράγματα. Να ρωτήσω ίσως την Κομισιόν. Αν πρέπει να ανησυχούμε ότι το θέμα αυτό μπορεί να γίνει επίμαχο και να κολλήσει αενάως στο Συμβούλιο. Υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο. Υποστήριζω πάντα στην έκθεση, είναι πολύ καλή, σωστή, αλλά πρέπει να ανησυχούμε για το τι θα συμβεί με το σημείο αυτό στο, στο Συμβούλιο. Μπορεί να απαντήσει η Κομισιόν. Για την Κομισιόν μπορούμε να απαντήσουμε, για το λογαριασμό τη Κομισιόν. Ε, το Συμβούλιο θα απαντήσει για το λογαριασμό του, για τι δικέ του εσωτερικέ διαδικασίε. Η Κομισιόν πιστεύει ότι η, οδηγία, η κατεύθυνση του εισηγητή είναι πολύ επικοδομητική και πρότεινε συμβιβασμό σε ό,τι αφορά την νομική βάση. Αυτή την έννοια δεν νομίζω λοιπόν ότι θα υπάρξει τεράστιο χάσμα ανάμεσα στο, στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο. Εμείς είμαστε έτοιμοι και στο σημείο αυτό να κάνουμε τα βήματα και σε ό,τι αφορά την προθεσμία για την επικύρωση που έχει παραταθεί, όπως πρότεινε και ο εισηγητής. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την Κομισιόν, η Κομισιόν μπορώ να σας πω ότι είναι έτοιμη να προβεί σε περαιτέρω διάλογο. Υποστηρίζουμε την επικύρωση των συντομότερων δυνατών, αλλά από όλα τα κράτη-μέλη. το συμφέρον της Ένωση. και να μην, δεν θέλουμε να κινηθούμε ανεξάρτητα ημένα του δε και κατακαιρματισμένα. Δυστυχώ, το Συμβούλιο δεν εκπροσωπείται στη συνεδρίαση, παρότι τους προσκαλέσαμε μία διόρθωση. Στην αγγλική μετάφραση γράφεται ότι η προθεσμία για τροπολογίες είναι 27 Μαΐου, ενώ το τσεχικό κείμενο, ε, που είναι και το, το πρωτότυπο, είναι, λέει, Απρίλιος 27 του μηνός, 27 Απριλίου δηλαδή, που είναι και η σωστή η ημερομηνία. Άρα, Κλείνουμε το σημείο αυτό και θα ξαναρχίσουμε στις 9.30 με ψηφοφορίες. Uh, Mrs. Boutonnet wishes to, to say something. Allez-y. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για μια αναβολή ψηφοφορίας. Καταρχάς, για το άρθρο 257 ε, ε, και ε, δεν υπάρχει καμία νομική βάση. Ε, και στο, στην στο σημείωμα τη νομική υπηρεσία δεν λέγεται τίποτα. Η κυρία Ντελβό μετά από τη συζήτηση τη προηγούμενη συνεδρίασης είχε ζητήσει μια λεπτομερή ανάλυση από την νομική υπηρεσία. Έχετε αναλύσει τι προπαρασκευαστικές εργασίες τη συνθήκη τη ε, Λισαβόνα, Νίκαια, είπε η ομιλήτρια. Την ομολογία του δικαστηρίου επίση, για παρόμοιε διατάξει. όχι. Ε, δεν έγινε καμία ε, μελέτη αντικτύπου για την μεταρρύθμιση του δικαστηρίου και επίσης για την ε, ε, κατάργηση του δικαστηρίου και το κόστος. Ούτε για το διπλασιασμό του αριθμού των δικαστών. Υπάρχει ένα μεγάλο άρθρο ε, που δημοσίευσε ένας δικαστής στο δικαστήριο, το οποίο είναι πολύ έγκυρο. Ο συντάκτης έχει σκεφτεί μέτρα εξορθολογισμού που ε, αύξαν πάρα πολύ τις υποθέσεις που έκλεισαν, μειώθηκαν πάρα πολύ α, οι χρόνοι διεκπαιρέωσης μιας υπόθεσης. Αυτό το άρθρο που είναι πολύ επτομερές δείχνει πως αυτή η μη απαραίτητη μεταρρύθμιση έγινε ε, παρά τα όσα επιτάσσει λογική. Υπάρχει θέμα. Ε, αυτή η μεταρρύθμιση ε, επιδίνωσε την εικόνα του δικαστηρίου, ε, του, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ε, ο συνάδελφος Μάριο Πίντο ε, είπε κάποια πράγματα, αλλά τον αγνοήσατε. Υπάρχουν άλλες λύσεις από το διπλασιασμό των δικαστών, πολύ πιο αποτελεσματικός. Ε, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Θα πρέπει να δούμε τα πράγματα με κάποια απόσταση ε, τη στιγμή που σε όλα τα κράτη υπάρχει η λογική της λιτότητας. Επομένως, θέλω να καθυστερήσουμε αυτή τη ψηφοφορία, να διαβάσετε αυτό το άρθρο του καθηγητή Φρόνκλεον de και να ε, φτάσετε στα σωστά συμπεράσματα. Επίσης, θα πρέπει οι κλητήρες του δικαστηρίου να έρθουν εδώ και να, σε μια ακρόαση κτλ. Ε, καθώς και οι δικαστές. Αλλιώς μπορούμε να πούμε ότι αυτή η Επιτροπή ε, λειτουργεί εν απουσία δικαίου. Ευχαριστώ πολύ για την ε, ένσταση και την ανάλυση. Άρα πρέπει να ε, ψηφίσουμε το αν θα γίνει ψηφοφορία, αφού έχετε αμφιβολίες. Παρακαλώ τους αγαπητούς συναδέλφους να συγκεντρωθούν εδώ. Εννέα και 30 θα ξεκινήσει η προφορία τους ή άλλως. Άρα ξανά ανακοινώνω το διάλειμμα. 9 και 30 για να είναι παρόντες όσοι θα το επιθυμούσαν. Euh, Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινώ. Είναι 9 και 31. Και πριν ξεκινήσουμε παρακαλώ να βεβαιωθείτε πως έχετε τις ε, κάρτες για την ψηφοφορία. Είστε όλοι εξοπλισμένοι. Άριστα. Λοιπόν, ακούσατε την έσταση ε, της συναδέλφου. για όποιον δεν ήταν μέσα στην αίθουσα, υπενθυμίζω ότι η συνάδελφος ζήτησε την αναβολή της ψηφοφορία για την ε, παραπομπή στο δικαστήριο. Έχετε πρόβλημα, δεν έχετε κάρτα. Καλά, θα σας κοιτάμε τότε, εντάξει. Θα έχετε την αμέριστη προσοχή της γραμματείας σήμερα. Λοιπόν, ερωτώ αγαπητοί φίλοι, εάν υπάρχουν ε, αντιρρήσεις στην επιχειρηματολογία της συναδέλφου που ζήτησε την αναβολή. Καλώς λοιπόν. Θα ψηφίσουμε αυτό το ζήτημα λοιπόν. Ποιος θέλει να παραμείνει η στην ημερήσια διάταξη ψηφοφορία. Σηκώστε τα χέρια σας παρακαλώ για να μπορώ να μετρήσω. Τέσσερις. Δεκατρεις υπέρ. Αποχές λέει ο πρόεδρος. Μία αποχή. Κατά. Κατά της διατήρησης της ψηφοφορίας. Και ο κύριος Τζεμπάτσκι, τρεις. Το όλον. 13 υπέρ, 3 κατά μία αποχή. Ψηφοφορία λοιπόν θα λάβει χώρα ευθύς αμέσως και ξεκινώ με την ψηφοφορία. Τροπολογίες 2, 3, 4 υπέρ. 2, 3, 4 υπέρ. Δεν χρειάζεται να μετράω. Κατά. Αποχές. Και εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ. Αποχές και κατά. 7 υπέρ. Αποχές. Κατά. Και απορρίπτεται. 8 υπέρ. Αποχές. Κατά. Απερίφθη. 9 Υπεραποχές κατά Απερίφθη το σύνολο τώρα της εκθέσεως όπως τελετήθηκε ηλεκτρονικά αρχίζει η ψηφοφορία Έχω ένα μικρό πρόβλημα και εγώ με την ε, κάρτα μου. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, αν δεν έχετε αντίρρηση, σας παρακαλώ να ξαναρχίσει αυτή η ηλεκτρονική ψηφοφορία, να την επαναλάβουμε, γιατί δεν λειτουργεί σωστά το σύστημα. Άρχεται η ψηφοφορία. Αποτελέσματα. 15 υπέρ. 4 κατά. Αποχή ουδεμία. Και έτσι εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Αποχές. Κατά. Απερίφθη. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές μάλλον. Αποχές και κατά. Απερίφθη. Ονομαστικά το ψήφισμα. Ηλεκτρονικά. Πέρας. 16 υπέρ. 4 κατά εγκρίνεται. Ηλεκτρονικά εντολή διαπραγματεύσεων. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 17 υπέρ, 3 κατά και συγχαρητήρια. Τώρα ψηφίζουμε την νομική βάση Et on va le faire à celui celui-là. Il a pas Και τώρα η ψηφοφορία της ε, ε του κύριου Φως, ο οποίος το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ στο υπόμνημα για τη μεταφορά στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο και τις τροποποιήσεις που θα προκύψουν σε σχέση με το δικαστήριο για τους υπαλλήλου θα θέλαμε να διαγραφούν στο, από το υπόμνημα αυτό την νομική πραγματογνωμοσύνη δύο φράσεις. Αν μου επιτρέπετε πολύ σύντομα να τις παρουσιάσω. Τελευταία φράση της σελίδα 4, εκεί όπου λέγεται ότι πρόκειται για ένα άρθρο της ε, συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν καλύπτει την περίπτωση καθώς ε, δεν ε, επιτρέπει την λήψη συγκεκριμένου τύπου αποφάσεων με την μεταβίβαση των εξουσιών. Και αυτό πρέπει να διαγραφεί όπως και στη σελίδα 5 στο δεύτερο, στη δεύτερη τελεία, τελευταία φράση πάλι, εκεί που λέει να μην ορίζεται ότι όλα τα, όλες οι λειτουργίες του δικαστηρίου πρέπει να έχουν την ευλογία του αιωνίου φωτός. Συμφωνώ λοιπόν με την πρόταση να διαγραφούν οι δύο αυτές φράσεις. Και ακόμα και αυτή σχετική με το αιώνιο φως, με το άσβεστο φως.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 την εκθέση της κυρίας Χάουταλα. Σχόλιο. Κύριε Χάουταλα. Ναι, Πρόεδρε, μου δίνετε το λόγο για πολύ λίγο. Θα ήθελα να εξηγήσω κάποιες μικροαλλαγές από την ομάδα εργασίας για το διοικητικό δίκαιο από την ε, πρώτη παρουσίαση αυτής της πρότασης στην Επιτροπή μας. Ξέρετε ότι στόχος της πρότασης ήταν ε, να καταστεί προς παράρτημα στο ψήφισμα ε, κατόπιν της επί της προφορικής ερωτήσεως με... και έχουμε τίτλο «Ανοιχτή αποτελεσματική και ανεξάρτητη Ευρωπαϊ... διοίκηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση». Αποφάσισε λοιπόν η ομάδα εργασίας νέο τίτλο για το κείμενο της πρότασης ώστε να αντιστοιχεί και στην νομική βάση, δηλαδή το άρθρο 298 για την, τις συνθήκες για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέος τίτλος λοιπόν, πρόταση κανονισμού για ανοιχτή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη διοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθαρά δηλαδή γλωσσική προσαρμογή και Έχοντας υπόψη και τα σχόλια του κυρίου Σκουρή, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην ακρόαση τον ε, Ιανουάριο, αποφασίσαμε για τα ένδικα μέσα στο άρθρο 20 να κάνουμε μια μικροδιόρθωση για να διευκρινιστεί και η δυνατότητα αξιοποίησης της διοικητικής προσφυγής και αναθεώρησης, η οποία δεν θα παρεμποδίσει, δεν θα οδηγεί δηλαδή σε εκπνοή των προθεσμιών για την υποβολή προσφυγής στη συνέχεια στο δικαστήριο. Έτσι λοιπόν γίνεται η σχετική προσαρμογή και τα κείμενα παίρνουν αριθμό οι παράγραφοι 33 και 34 αντίστοιχα. Έτσι πιστεύω μπορούμε να πάμε με την υπόθεση αυτή, δείχνοντας ότι ως Κοινοβούλιο έχουμε αντιληφθεί πως πρόκειται για μια μακρά διαδικασία και αυτό ως δώρο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ψηφοφορία λοιπόν για την προφορική ερώτηση πρώτα και μετά το ψήφισμα. Διανατάσσεως στην προφορική ερώτηση. Αποχές κατά. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται και τώρα το ψήφισμα υπέρ. Αποχές κατά. Ευχαριστώ και εγκρίνεται. Κύριε Τζαμπάσκι, θέλατε το λόγο. Καλώς ευχαριστώ. Στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη πρόκειται για την έκθεση της κυρίας Ντελβό. Την ψηφίζουμε, θέλετε το λόγο όχι. Ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν. Αρχίζει. ηλεκτρονικά. Ευχαριστώ. Πέρας. 18 υπέρ, δύο κατά και εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Στο 22 τώρα στην ημερήσια διάταξη. Με ανάταση υπέρ κατά αποχές και εγκρίνεται 23 Έκθεση φως θέλετε το λόγο Όχι τον λάβατε ήδη σωστά Ψηφίζουμε διανατάσεως Αποχές κατά Κατά παρακαλώ τρεις ψήφοι κατά. Και εγκρίνεται. Και έτσι λοιπόν ε, εξαντλήσαμε τις οφορίες. Έχουμε μερικά λεπτά διάλειμμα μέχρι το επόμενο θέμα. Ένα τεταρτάκι λοιπόν διάλειμμα για την, μέχρι την ακρόαση στις 10.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

Όχι όχι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 Uh, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, καλημέρα σας. May we begin welcome. Να ξεκινήσουμε καλωσορίζοντας όλους τους παριστάμενους στην ακρόαση για τις νομικές και ηθικές διαστάσεις της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης. Να καλωσορίσω τους προσκεκλημένους μας. Θα τους ε, παρουσιάζω καθώς θα παίρνουν το λόγο. Καλωσορίζω και την ε, συνάδελφο Μαγκλέν Τελβό που είναι υπεύθυνη για την ομάδα εργασίας για την νομοθεσία για τη ρομποτική. Και επειδή η καθηγήτρια Βέντεχος, η πρώτη μας προσκεκλημένη, θα πρέπει να φύγει σύντομα, θα ξεκινήσουμε αμέσως. Οπότε δίνω το λόγο στην Κριστιάνε Βέντεχος, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Βιέννης, να μας μιλήσει για την ρομποτική, την τεχνητή νοημοσύνη και τις συμβάσεις μεταξύ μηχανών. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε σε αυτήν την ακρόαση. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ. Ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη και συμβάσεις μεταξύ μηχανών είναι ένα τεράστιο θέμα βεβαίως. Θα μπορούσα να μιλήσω ώρες, οπότε με την άδειά σας, επειδή χρειάστηκε να κάνω μια επιλογή, θα επικεντρωθώ σε κάποια ζητήματα που υποθέτω ότι δεν θα, τις καλύψουν, δεν θα τα καλύψουν οι επόμενες ε, παρουσιάσεις, συγκεκριμένα στις συμβάσεις καταναλωτών. Πρώτον, τι είναι ακριβώς μια σύμβαση μεταξύ μηχανών. Όπως γνωρίζετε, η ισχύουσα νομοθεσία δεν αποδίδει νομική προσωπικότητα σε μηχανήματα. Άρα, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί η νομοθεσία να εννοεί ε, συμβάσεις που ε, συνάπτονται μεταξύ δύο μηχανημάτων, δηλαδή μιας μηχανής αγοραστή και μιας μηχανής πολιτή. Άρα πρέπει να σημαίνει ε, κάτι άλλο. Ας εξετάσουμε λοιπόν κάποια σενάρια. Σενάριο 1. Η Κάρολ διαβάζει κάποιες σελίδες στο online shop του Bill και μόλις διαπιστώνει ότι η αγαπημένη της σαμπάνια προσφέρεται σε μια πολύ καλή τιμή, συμπληρώνει μια ηλεκτρονική φόρμα και κάνει την παραγγελία της. Η παραγγελία αυτή παραλαμβάνεται από το αυτοματοποιημένο σύστημα επεξεργασίας παραγγελιών του Bill, το οποίο ελέγχει αν υπάρχουν στο απόθεμα τα μπουκάλια της σαμπάνιας και στέλνει μια ε, επιβεβαίωση στο email της Κάρολ. Πρόκειται για μια ε, σύμβαση μεταξύ μηχανωμάτων, προφανώς όχι. Πρόκειται για μια ε, συναλλαγή ηλεκτρονικού εμπορίου διότι το κρίσιμο βήμα, δηλαδή η πραγματοποίηση της παραγγελίας, έγινε με ανθρώπινη παρέμβαση. Φυσικά, όλα τα προβλήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως για παράδειγμα το πώς θα μπορούσαμε να διασφαλίσουμε ότι πραγματικά η Κάρολα έκανε αυτή την παραγγελία, πώς θα διασφαλίσει κανείς ότι το, την ακαιρεότητα του μηνύματος και ότι κανείς δεν παρεμβλήθη ε, κατά τη διαδικασία διαβίβασης της ε, παραγγελίας. Όλα αυτά αφορούν βεβαίως την προστασία των δεδομένων. Αλλά εδώ μιλάμε για μια κλασική περίπτωση ηλεκτρονικής συναλλαγής, ηλεκτρονικού εμπορίου δηλαδή δεν εμπλέκονται μηχανήματα. Α πάμε όμω σε ένα, ένα βήμα παραπέρα, Α δούμε ένα δεύτερο σενάριο. Η Κάρολ ε, αγαπάει πολύ του υπολογιστέ υπολογιστές και προγραμματίζει τον υπολογιστή του ώστε να παρακολουθεί τι τιμέ στο online shop του Bill. Και μόλι κάποια στιγμή η σαμπάνια πέσει, η τιμή τη σαμπάνια, δηλαδή πέσει κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο που έχει θέσει η Κάρολ, ο υπολογιστή τη αυτόματα κάνει μια παραγγελία για αυτά τα 12 μπουκάλια σαμπάνια και ε, η παραγγελία αυτή παραλαμβάνεται από το σύστημα επεξεργασίας παραγγελιών του Bill. Αυτό είναι ένα πολύ απλό μοντέλο σύμβασης M2M μεταξύ μηχανών, διότι το βασικό, το κρίσιμο βήμα δεν γίνεται μέσω ανθρώπινης παρέμβασης, αλλά έμεσα μέσω της του προγραμματισμού ενός αλγορίθμου. Άρα το, η παρακίνηση για να πραγματοποιηθεί αυτή η παραγγελία έγινε από μηχάνημα έπειτα από ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο ε, διαπίστωση στοιχείων, σχεδιασμού και δράσης. Αλλά εδώ δεν μιλάμε μόνο ε, για, ε, για, αυτά τα, για αυτού του είδους τις συμβάσεις. Μιλάμε για δισεκατομμύρια ευρώ που θα συναλλάσσονται τα επόμενα χρόνια μεταξύ μηχανημάτων. Εδώ όμως δεν μιλάμε για ανθρώπους που αγαπούν απλά τους υπολογιστές και ξέρουν να προγραμματίζουν. Μάλλον θα συμβαίνει το εξή. Σενάριο 3. Η Κάρολ έχει αγοράσει ένα έξυπνο ψυγείο, το οποίο ε, το έχει πουλήσει η Σάλη και το οποίο το έχει κατασκευάσει ο Πολ, το οποίο αυτόματα παρακολουθεί το απόθεμα και στη συνέχεια κάνει τα ψώνια ε, σύμφωνα με ορισμένες προδιαγραφές και στοιχεία που η Κάρολ έχει ορίσει. Όταν λοιπόν η σαμπάνια στο ψυγείο της Κάρολ πέσει κάτω από μια συγκεκριμένη ποσότητα οριστήσα, το λογισμικό αγορών ε, αναζητεί κατευθείαν πρόσφορες στο ίντερνετ, συγκρίνει τιμές και κάνει και την παραγγελία για τα νέα μπουκάλια. Αυτό αυτή η παραγγελία μετά παραλαμβάνεται από ένα σύστημα επεξεργασίας παραγγελιών. Αυτό δεν αφορά μόνο ψυγεία, αφορά και τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα που μπορούν να παραγγέλνουν ανταλλακτικά αυτόματα και υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για τις επιχειρήσεις σε αυτόν τον τομέα. Αυτό λοιπόν είναι μια πρότυπη περίπτωση σύμβασης M2M περιλαμβάνει τουλάχιστον τρία συμβαλόμενα μέρη. Υπάρχει ο ιδιοκτήτης του μηχανήματος, ο ε, παραγωγός ή προγραμματιστής του μηχανήματος και φυσικά υπάρχει και το συμβαλόμενο τρίτο μέρος, συν ε, τυχόν ε, πολιτές, ενδιαμέσους, εμπόρους, ε, παραγωγούς άλλων μηχανημάτων κτλ. κτλ. Μπορεί να υπάρχει μια σύμβαση πλαίσιο μεταξύ του C και του B ε, για παράδειγμα το υποκατάστημα μιας αλυσίδας ε, ε, τροφίμων που λειτουργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ του C και B που στην πραγματικότητα κάνουν μεταξύ τους αυτή τη συναλλαγή ή μπορεί να υπάρχει και μια ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία διαμεσολαβεί και οργανώνει αυτές τις συναλλαγές σε ευρύτερη κλίμακα. Όλα αυτά τα ζητήματα ε, τα ρυθμίζει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Να δούμε την ε, οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Εκεί υπάρχουν κάποιες προσυμβατικές πληροφορίες, αλλά αυτές οι πληροφορίες καταλήγουν στο ψυγείο. Δίνονται στο ψυγείο. Αν δούμε την μεμονωμένη ε, συναλλαγή. Αυτό έχει συμβεί και το ίδιο ισχύει και σε άλλες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, όσον αφορά την, την ε, των ε, σφαλμάτων καταχώρησης. Αν δούμε πάλι την οδηγία για τα δικαιώματα του καταναλωτή, εκεί δεν έχει ε, συνταχθεί η οδηγία αυτή έχοντας κατά νου ε, τις συμβάσεις M2M ε, γιατί δεν προβλέπεται να δίνονται πληροφορίες σε μηχανήματα ούτε ε, υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις προβλέψεις όσον αφορά τις απαιτήσει για τις επιβεβαιώσεις, την επισήμαση των κουμπιών κτλ. Η οδηγία για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές και τους αθέμητους όρους τους, αν συμβατικούς όρους, ε, αφήνει στα κράτη-μέλη να ρυθμίσουν ε, τα ζητήματα αυτά και κατ' επέκταση και τις ε, συμβάσεις M2M. Για παράδειγμα, τι συμβαίνει όταν υπάρχει ε, από τη μία πλευρά ένας άνθρωπος, μια συναλλαγή δηλαδή, και από την άλλη ένα ψυγείο. Τι συμβαίνει αν τα πράγματα πάνε άσχημα και ποιος, σε πάση περιπτώσει, αναλαμβάνει την ευθύνη. Ας δούμε λοιπόν την οδηγία για την ε, ευθύνη για τα ελωτηματικά προϊόντα. Εδώ δεν καλύπτονται οι καθαρές οικονομικές απώλειες και στην, ε, ε στις ε, συμβάσεις μεταξύ μηχανημάτων συνήθως για κάτι τέτοιο μιλούμε, δεν, δεν μιλούμε για τραυματισμούς ας πούμε. Αν δούμε την οδηγία για τις πωλήσει καταναλωτών θα πρέπει να πούμε αν η, ο καταναλωτής Κάρολ έχει οποιασδήποτε δυνατότητες προσφυγής ανάλογα με κάποιους παράγοντες. Για παράδειγμα, αν, ε, το, το σφάλμα, αν το σφάλμα έγινε από την ίδια την Κάρολ ή αν ε, το ε, μηχάνημα δεν λειτουργήσε με βάση τους συμβατικούς όρους. Ποιος λοιπόν ε, βαρύνεται με αυτήν την ευθύνη. Αλλά κυρίως η συγκεκριμένη οδηγία δεν ε, προβλέπει δικαίωμα αποζημιώσεων, αυτό ε, εναποτίθεται στις εθνικές νομοθεσίες. Και εκεί μπορεί και να προβλέπεται υποχρέωση απόδειξης ευθύνης. Αν δούμε την, ε, το σχέδιο οδηγίας για τις συμβάσεις για την παροχή ψηφιακού περιεχομένου, εδώ δεν καλύπτονται λογισμικά που είναι ενσωματωμένα σε φυσικά αγαθά, καλύπτει την παροχή, την παροχή συγκεκριμένων πρακτόρων λογισμικού, αλλά τα, οι έλεγχοι ε, συμμόρφωσης αφορούν και ενσωματώνονται στους όρους και τις προϋποθέσεις. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι στις συμβάσεις M2M οι συνήθεις εγγύησεις για την εξασφάλιση μιας αυτόνομης λήψης απόφασης μπορεί να ε, μην αφορά τελικά την ίδια την συναλλαγή. Ο κάτοχος, ο ιδιοκτήτης, κάνει αυτόνομες συμβατικές αποφασίσεις, αλλά μόνο ε, νωρίτερα στον χρόνο και συγκεκριμένα όταν υπογράφει μια σύμβαση πλαίσιο είτε άμεσα με τον αντισυμβαλόμενο ή με τον ενδιάμεσο που τον εκπροσωπεί και πολύ συχνά δεν υπάρχει ευθύνη των πολιτών ή των κατασκευαστών. Αν κάτι πάει άσχημα, για παράδειγμα, αν το έξυπνο αυτό ψυγείο ε, παραγγείλει υπερβολικά πολύ φαγητό ή αν κάποια στιγμή ένα smartphone ε, χρησιμοποιήσει online υπηρεσίες ε, ενώ ο ιδιοκτήτης είναι στο εξωτερικό. Ας πάμε και ένα, σε ένα επόμενο σενάριο, το σενάριο 4 που εδώ μιλούμε πραγματικά για τεχνητή νοημοσύνη. Ας φανταστούμε λοιπόν ότι η Κάρολ έχει αγοράσει ένα πολύ προηγμένο έξυπνο ψυγείο ε, το οποίο μπορεί να, με, με διάφορους αισθητήρε να σκανάρει το, το περιβάλλον του. Και ξέρετε ότι τα μηχανήματα μαθαίνουν με βάση την εμπειρία του μετά από κάποιους μήνες λοιπόν το ψυγείο γνωρίζει τα πάντα σχετικά με τις συνήθειες και προτιμήσεις της Κάρολ και αρχίζει και παίρνει αυτόνομες αποφάσεις λαμβάνοντας ε, υπόψη όλους αυτούς τους παράγοντες και τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του λαμβάνοντας υπόψη και βεβαίως τις προσυμβατικές πληροφορίες και τους όρους των ε, προμηθευτών του. Αυτό είναι πράγματι μια κανονική σύμβαση M2M. Ακριβώς γιατί περιλαμβάνει προηγμένη τεχνητή νομοθεσία. Τα ίδια τα άτομα, τα φυσικά πρόσωπα δεν παρεμβαίνουν σε μεγάλο βαθμό. Τι Νομικέ διαφορές υπάρχουν σε σχέση με το σενάριο 4. Λοιπόν, η προηγμένη ε, ε, τεχνητή νομιμοσύνη μπορεί να σημαίνει ότι μπορεί να συναπτονται συμβασει συμβάσεις M2M σε πολύ ευρύτατη κλίμακα και να μην ε, συνάπτονται μόνο εντό του πλαισίου των, των συμβάσεων πλαίσιο. Επίσης, αυτό όμως δημιουργεί μεγαλύτερου κινδύνους και κατά συνέπεια θα χρειαστεί να ε, καταρτιστεί και να θεσπιστεί νέα νομοθεσία και νέα ρυθμιστικά μοντέλα για όλα αυτά τα ζητήματα. Συνοψίζοντας, όταν εξετάζει κανείς ε, την σύναψη συμβάσεων M2M, ιδιαίτερα στον τομέα των καταναλωτών, πρόκειται για μια αγορά ε, που αναπτύσσεται ταχύτητα. Υπάρχουν πάρα πολλά μοντέλα, πρόκειται για συναλλαγές που συνάπτονται ή διενεργούνται εντός μιας σύμβασης πλαισίου συναλλαγές που πραγματοποιούνται εντός ορισμένων πλαισίων που έχουν, ε, ε, που έχουν θεσπίσει ενδιάμεση ή φορείς λειτουργίας πλατφορμών δηλαδή υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες ε, παράμετροι οι οποίοι έχουν καθοριστεί από τον κατασκευαστή σε συνεργασία με τον καταναλωτή και υπάρχουν και αυτόνομες συναλλαγές που ενδεχομένως να είναι το μέλλον όταν μιλούμε για προηγμένη τουλάχιστον τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρειαστεί περαιτέρω ε, νομοθετική ρύθμιση για να εξασφαλίζεται η δίκαιη κατανομή των κινδύνων, η, επαρκής, ε, η επάρκεια των πληροφοριών, η προστασία σε περιπτώσεις δυναμικής τιμολόγησης ε, για συναλλαγές M2M, μπορούμε να μάθουμε, για παράδειγμα, από τις υπηρεσίες πληρωμής σε αυτόν τον τομέα, οπότε πιστεύω ότι χρειάζεται περαιτέρω νομοθετική ε, ρύθμιση, ενώ οι ισχύοντες κανόνες αστικής ευθύνης για τη ζημία που προκαλείται στον κάτοχο ενός μηχανήματος ή σε τρίτους, στο πλαίσιο των ε, συμβάσεων M2M θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Αυτά λίγο χρόνο είχα δυστυχώς στη διάθεσή μου. Θα μπορούσα να πω πολύ περισσότερα για την τεχνητή νοημοσύνη και τις συμβάσεις M2M, αλλά δυστυχώς ε, ε, αυτά είχα το χρόνο να πω και βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Και μια και πρέπει να φύγει η καθηγητρία Χόστ. Ίσως θα ήταν τώρα η ώρα να ε, δεχθούμε τις ερωτήσεις προς αυτήν. Για τους λοιπούς ομιλητές θα ακούσουμε όλες τις ομιλίες και μετά. Λοιπόν, προς την ε, καθηγήτρια Πέντερφος υπάρχουν ερωτήσεις. Κύριε Ντελβού. Πρόεδρε, ευχαριστώ. για την ενδιαφέρουσα αυτή η παρουσίαση, Κριστίν. Βεβαίω έχω ερωτήσεις. Ίσως θα πρέπει, είπε, στο ενοχικό δίκαιο να αναθεωρηθεί το θέμα της ευθύνης ε, ε, έναντι τρίτων. Τι εννοείς ακριβώς δηλαδή. Θα πρέπει να αναγνωριστεί νομική προσωπικότητα στο μηχάνημα. Πώς το βλέπεις. Απάντηση. Εσείς ε, αναφέρεστε σε μια e-personality, ηλεκτρονική προσωπικότητα. Δεν μπόρεσα να επισέλθω σε λεπτομέρειες, δεν είχα αρκετό χρόνο, αλλά πιστεύω ότι για τα μοντέλα που μας αποσχολούν σε ευρεία κλίμακα και πάτησε ήταν οπωσδήποτε όχι. Υπάρχουν πολλά προβλήματα σε διάφορα επίπεδα. Φερρυπίν, πιθανή ανισότητα ε, στον επιμερισμό του κινδύνου σε συμβατικές σχέσεις, σε ενδιάμετα, ενδιάμεσα σχήματα όπου δεν υπάρχει επάρκεια ασφαλείας και προστασίας για τον μεμονωμένο καταναλωτή ο οποίος έχει ελάχιστο και καθόλου έλεγχο στο τι συμβαίνει, στο τι έχει επιλέξει ο προμηθευτής, στο πώς, κάνω, πώς γίνονται οι υπολογισμοί και ούτω καθεξής. Και έτσι, το να μιλήσουμε πιστεύω στο προκείμενο για ηλεκτρονική προσωπικότητα, νομική προσωπικότητα για τα μηχανήματα δηλαδή, δεν είναι ζήτημα. Φυσικά, αν κοιτάξουμε πιο μακριά, σε πιο προηγμένα μοντέλα σε συμβασει μεταξυ μεταξύ μηχανών, M2M contracting, όπου οι μηχανές μπορεί να είναι αυτόνομες όσο και ένας ε, δρόν άνθρωπος, τότε υπάρχει κενό ευθύνης, γιατί ο παραγωγός δεν έχει λόγω της οδηγίας περί παραγωγού ευθύνη, όπως έχει τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, οι αρμόδιοι για το χειρισμό πάλι δεν έχουν και έτσι αντιμετωπίζουμε κενό ως προς το τομέα της ευθύνης εδώ. Διάφορα μοντέλα υπάρχουν για το πώς μπορεί να κλείσει αυτό το κενό. Με δύο κύριους κλάδους ή σχολές, όπου η πρώτη σχολή θα έλεγε ότι μπορούμε να καλύψουμε το θέμα δημιουργώντας νέες κατηγορίες αστικής ευθύνης και μάλιστα αυστηρής περιγραφής και εκεί θα πρέπει να δούμε αν θα πρέπει να είναι κυρίως στον παραγωγό ή στον χρήστη και μετά βεβαίως θα πρέπει να ορίσουμε και υποχρεωτικά συστήματα ασφάλισης για αυτή την ευθύνη και αυτή τη σχολή ακολουθώ και εγώ ενώ υπάρχει μια άλλη σχολή που λέει ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί η έννοια του, της ηλεκτρονικής προσωπικότητας και να ε, προσλάβει ένα πολύ προηγμένο βέβαια μηχάνημα, νομική προσωπικότητα, να προσλάβει περιουσιακά στοιχεία και εάν προβαίνει σε σύμβαση που δεν είναι ικανοποιητική για το καταναλωτή ή ιδιοκτήτη, θα μπορεί ο καταναλωτής ή ιδιοκτήτης να κάνει αγωγή στο μηχάνημα, στη μηχανή ή και ο τρίτος αντισυμβαλόμενος θα μπορεί να κάνει τη σχετική αγωγή. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται αυτό γιατί προσθέτει επιπλέον περιπλοκές, δεν είναι απαραίτητο. Δεν νομίζω ότι επιτυγχάνει περισσότερα σαν αποτέλεσμα από ότι ένα πιο περίπλοκο σύστημα αστικής ευθύνης με υποχρεωτική ασφάλιση. Αυτό βλέπω εγώ. Νομίζω με αυστηρό σύστημα ευθύνη και ασφάλιση επιτυγχάνονται πολλά πράγματα και δεν μπορούν να επιτευχθούν περισσότερα, ε, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, ε, με την πρόσδοση νομικής προσωπικότητας. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κύριος Λεπρετό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την ε, καθηγήτρια για την παρουσίαση της εδώ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ σαφής. Κατέληξα και εγώ στις δύο συμπεράσματα ε, ακούγοντάς την. Θα τη συγχαρώ λοιπόν για άλλη μια φορά. Ε, περισσότερο παρά θα κάνω ερωτήσεις. Ιδιαίτερα το παράδειγμα του ψυγείου το οποίο είναι συνδεδεμένο και μπορεί να κάνει την παραγγελία ε, μερικών φιαλών σαμπάνιας όταν ε, τελειώσει αυτή. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα βέβαια. Υπάρχουν πέραν αυτού άλλα ζητήματα που έθιξε τώρα και η κυρία Ντελβό, το ζήτημα της ηλεκτρονικής προσωπικότητας που μου φαίνεται μάλλον επαναστατικό και ε, τρομακτικό, δηλαδή να δοθεί ευθύνη σε μηχανή και να μπορεί κανείς να κάνει αγωγή κατά μιας μηχανής και βεβαίως Η άλλη λύση θα ήταν μια ευθύνη του παραγωγού ή του ιδιοκτήτη κατά, κατά περίπτωση, ανάλογα με την φύση του προβλήματος και υποχρεωτική ασφάλιση ε, αστικής ευθύνης. Αυτή νομίζω ότι είναι η πιο λογική ευθύνη και με χαρά ακούω ότι μας προτείνει αυτό και η καθηγήτρια Βέντερχορστ σήμερα. Και πάλι ευχαριστώ για την πολύ καλή παρουσίαση. Η καθηγήτρια Βέντερχορστ θα ήθελε να αντιδράσει ή δεν νομίζω. Ευχαριστώ. Όπως σας είπα, το θέμα της ευθύνης είναι ένα θέμα που άπτεται όλων των υπόλοιπων θεμάτων που μας απασχολούν. Είναι κάτι το οποίο Αφορά και το, τη συμβατική σφαίρα, αλλά και την έξω συμβατική σφαίρα. Όταν ένα ρομπότ, ας πούμε, προκαλεί φυσική βλάβη ή καταστροφή. Είναι ένα διατομιακό θέμα, θα έλεγα. Και εγώ προσωπικά θεωρώ ότι δεν χρειαζόμαστε αυτή την ε, νομική προσωπικότητα. Πρέπει να σκεφτούμε αυστηρή ευθύνη και κάποιο έτσι περίπλοκο και πολύ καλό σύστημα ασφάλισης. Πέρα, από αυτή, πέρα και κάτω από αυτή τη συζήτηση και το, την πολύ επαναστατική ιδέα της, ε, της ε, ηλεκτρονικής ε, προσωπικότητας υπάρχουν διάφορα άλλα θέματα πιο παραδοσιακά που μπορούμε να τα ξεχάσουμε. Παραδοσιακά προβλήματα για τις αυτόνομες αποφάσεις, για τους όρους της σύμβασης, για τα μοντέλα τιμολόγησης, για το δίκαιο ανταγωνισμού. Υπάρχει κάποιος ενδιάμεσος συνήθως, ο οποίος αποφασίζει ποιος θεωρείται προμηθευτής και ποιος δεν μπορεί να θεωρηθεί προμηθευτής και που διαπραγματεύεται, ας πούμε, έτσι, στα μετόπιστε, να πούμε, αν θέλετε, τις ε, τιμές που τελικά θα πρέπει να πληρώσουν οι καταναλωτές. Και θα ήθελα να τονίσω το εξή ότι η όλη συζήτηση για την ε, ηλεκτρονική προσωπικότητα και τα συστήματα ευθύνη είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πολλά μπανάλ, παραδοσιακά προβλήματα ε, που αφορούν τη συμβατική σφαίρα, το δίκαιο του ανταγωνισμού και που θα πρέπει ίσως να εξετάσουμε και να είμαστε σίγουροι ούτως ώστε ε, να είμαστε σίγουροι ότι οι καταναλωτές ε, απολάβουν επαρκούς προστασίας. Η κυρία Κομοντίνη. Καταλαβαίνω, εστιάζουμε πιο πολύ στην υπόθεση ε, της φυσικής ε, ζημίας. Ε, όταν μιλάμε για μηχανήματα που μπορούν να μάθουν και που συνδέονται μεταξύ τους, τότε θα πρέπει να δούμε τις συνήθειες του ιδιοκτήτη, της οικογένειας στην οποία βρίσκονται, και επίση μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ε, μηχανέ που έχουν το δυναμικό να παραγγέλνουν ας πούμε μπουκάλια ε, σαμπάνιας από ένα ε, ψηφιακό μαγαζί. Έχουν όλα αυτά τα προσωπικά δεδομένα σου λοιπόν και μην ξεχνάτε ότι μπορεί το μηχάνημα να αποκαλύψει τα προσωπικά σου δεδομένα. Θα πρέπει να σκεφτούμε και την ευθύνη σε αυτή την περίπτωση. Μιλάμε για την ίδια την κυρίως ηλική ζημία που μπορεί να επιφέρει η μηχανή στο, στον άνθρωπο, αλλά υπάρχουν και θέματα ιδιωτικής σφαίρας που δεν θα πρέπει να τα ξεχνάμε. Well, absolutely. Προφανώς, λέει η καθηγήτρια. Δεν υπάρχουν ειδικά προβλήματα που έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουν να κάνουν... Η τεχνητή νοημοσύνη έχει να κάνει με τα πάντα. Ακόμα και χωρίς σύμβαση. Ακόμα και χωρίς ρομπότ. Χωρίς τεχνητή νοημοσύνη υπάρχουν έξυπνε συσκευέ γύρω μας. Με τεράστιο δυναμικό. Αποκάλυψης των προσωπικών μας ε, δεδομένων και εισβολή στην ε, ιδιωτικότητά μας. Είναι απόλυτα αληθές ότι πρέπει να βρούμε κάποια λύση ε, και γι' αυτό που δεν θα είναι και εύκολο να βρεθεί βεβαίω. Έχει να κάνει με το ότι υπάρχει διασύνδεση στα πράγματα. Ότι έχουμε άπειρες τεχνολογικές ε, δυνατότητες σήμερα. Και δεν συνδέεται κατά ανάγκη με την τεχνητή νοημοσύνη ή τις, σύμβασ, τις συμβάσεις μεταξύ μηχανημάτων. Φυσικά, ε, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επιτείνει το πρόβλημα, αλλά το πρόβλημα προϋπάρχει. Κύριε Κύριε Ντελβό. Μετά από αυτά που μας είπατε, το θέμα είναι ποιος ε, είναι ο ιδιοκτήτης των δεδομένων σε αυτές τις συμβάσεις μηχανή προς μηχανή ή για την πληρωμή των υπηρεσιών. Μπορείς να πληρώσεις με χρήμα ε, ή με δεδομένα. Τι γίνεται όλα αυτά, πώς εντάσσονται στο θέμα των συμβάσεων, δηλαδή τι πρέπει να μας απασχολήσει μιλώντας για τις συμβάσεις. Το να πληρώνεις με δεδομένα και ε, το θέμα της ιδιοκτησίας των δεδομένων, της κυριότητας των δεδομένων. Δεν έχει να κάνει μόνο με τις συμβάσεις. Έχει να κάνει με την επικοινωνία. Παραδείγματος, έχω ένα συνδεδεμένο αυτοκίνητο, το οποίο παράγει δεδομένα, τα οποία συνεχεία διαβιβάζονται σε τρίτους. Δεν χρειάζεται να υπάρχει σύμβαση εκεί στη μέση. το αυτοκίνητό μου δεν συνάπτει σύμβαση. Μιλάμε για επικοινωνία, μιλάμε για μεταβίβαση δεδομένων στην πραγματικότητα εδώ. Το να πληρώνεις με δεδομένα και το θέμα της κυριότητας των δεδομένων είναι κάτι που προσπαθεί η Κομισιόν να εξετάσει στην πρόταση για, τις, για την σύμβαση για την παροχή ψηφιακού περιεχομένου και εκεί έχει την προσέγγιση ότι οι συμβάσεις όπου πληρώνεις για το ψηφιακό περιεχόμενο με ειδικά προσωπικά δεδομένα έχουν την ίδια ε, σημασία με τις συμβάσεις ε, όπου πληρώνεις για το ψηφιακό περιεχόμενο με χρήμα. Εγώ πιστεύω ότι είναι σωστό αυτό. Βήμα προς σωστή κατεύθυνση είναι αυτό. Μην ξεχνάμε ότι μπορεί να θεωρηθούν τα δεδομένα ένα είδος νομίσματος. Μην ξεχνάμε όμως το εξής. Όταν εξετάζουμε δεδομένα, ή μάλλον όταν βλέπουμε ως νόμισμα, όταν τα βλέπουμε ως ένα είδος αντιτίμου, ως μια μορφή πληρωμής, όπου ο καταναλωτής ή ο αγοραστής ε, δίνει για να πάρει μια υπηρεσία ή αγαθά, τότε μπορεί να δυσκολεύσει η αγαθα τοτε μπορει να δυσκολέψει η σχεση ε, με το δίκαιο ε, προστασίας των δεδομένων. Γιατί εκεί το θέμα ε, του δικαιώματος που έχουμε να αποσύρουμε το, τη συνένεσή μας για την επεξεργασία των προσωπικών μας δεδομένων πάντα θεωρούς, θεωρεί πυλώνας του δικαίου αυτού προστασίας των δεδομένων. Και πάντα η άποψη υπερίσχυε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπάρχει καμία παρέκκληση από, την, από το δικαίωμα να αποσύρεις τη συνένεσή σου. Τώρα, αν το δούμε από διαφορετική όμως σκοπιά, αν θεωρήσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα είναι αντίτιμο, είναι πληρωμή, και αν μιλάμε για την κυριότητα των δεδομένων σαν κάτι ε, σαν ένα δικαίωμα, ας πούμε, πνευματικής ιδιοκτησίας που μπορεί να, το, να μπει σε συναλλαγή, ας πούμε, τότε αλλάζει η σχέση μας ε, με τα δικαιώματα που έχουμε, το δικαίωμα παραδείγματος χάρη να αποσύρουμε, ας πούμε, τη συγκατάθεσή μας για επεξεργασία των δεδομένων μας. Και μπορεί όλη αυτή η συζήτηση για την κυριότητα των δεδομένων ε, να μοιάζει σαν να δίνουμε περισσότερα δικαιώματα στο άτομο και να είναι το υποκείμενο ας πούμε και να βρίσκεται αυτό, και αυτό να κουμαντάρει την όλη ιστορία και μπορεί να είναι σωστό σε κάποιο βαθμό αλλά μπορεί να έχει και εντελώ αντίθετα αποτελέσματα. Μπορεί δηλαδή έμεσα, εάν σκεφτούμε όλες τις επιπτώσεις, να αποστερήσουμε το άτομο από το δικαίωμά του να αποσύρει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Εάν αν ξαφνικά τα δίνει αυτά τα δεδομένα, ας πούμε, ως αντίτιμο. Τότε το δικαίωμά του να αποσύρει τη συνένεσή του, τη συγκατάθεσή του, μπορεί να μην ε, συμβαδίζει με αυτή τη νέα προσέγγιση. Επομένω, να, να και ένα μειονέκτημα σε αυτή την ιστορία. Ευχαριστώ πολύ, καθηγήτρια Βέντερχορστ, που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ και για τις απαντήσεις σας. Δεύτερη προσκεκλημένη, δεύτερος προσκεκλημένος, ο κ. Παύλ Κριατκόφσκι από την ε, το νομικό γραφείο Γκέσελο της Βαρσοβίας. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ενοχικό δίκαιο και αδικοπραξία. Και ευθύνη μάλλον. Ξέρετε, Έχω έρθει σήμερα εδώ, Πρόεδρε, να σας δώσω ένα πυρουλάχιστο κομμάτι του ενοχικού δικαίου και του δικαίου της ευθύνης ε, σε σχέση με την ρομποτική. Αλλά μια και έχω μια ανταγωνιστικότητα χαρακτήρας, ε, θέλησα να σας δώσω ένα κομμάτι από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Το θέμα που θέλω να επισημάνω είναι ότι έχουμε να κάνουμε ζητήματα του αστικού δικαίου. Ένα κομμάτι του δικαίου που έχει πληρέστατη κάλυψη και έχει πει κάποτε ο καθηγητής μου ότι καλύπτει κάθε ε, παραμικρή δραστηριότητα ανθρώπου. Είτε αγοράζει εισιτήριο, είτε αγοράζει ε, κουστούμι, βρίσκεσαι πάντα μέσα στο πλαίσιο κάποιων διατάξεων του αστικού δικαίου. Με άλλα λόγια, δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα ζητήματα που μας απασχολούν εδώ, το αστικό δίκαιο δηλαδή, όπως έλεγε ένα παλιό τραγούδι για την αγάπη, είναι γύρω μας. Love is all around us. Με αυτά λοιπόν προχωρώ στο κύριο θέμα μου, την ε, αστική ευθύνη λοιπόν στην περίπτωση της ρομποτικής. Και πριν από την ε, συνεδρίαση εδώ έχω την ευκαιρία να συζητήσω ζητήματα αλλαγών στο πολωνικό σύστημα δικαίου και ε, συστήματα ανταλλαγών υψηλής ή συναλλαγών υψηλής ε, συχνότητας ή ταχύτητας στα χρηματιστήρια που μου επισημάνθησαν μάλιστα από έναν ειδικό εκεί στις συζητήσεις και γι' αυτό θα ήθελα να έρθω να σας τα αναφέρω και εσάς. Η high frequency trading, ε, συναλλαγές υψηλής ταχύτητας ψηκλής συχνότητα που ήδη συμβαίνει συμβαίνουν σήμερα. Δηλαδή δεν έχουμε να κάνουμε κάτι το μελλοντικό, αλλά μια πραγματικότητα. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό. Υπάρχει ένα σύστημα αλγορίθμων για τις ε, αγοραπολισίες σε επίπεδο χρηματιστηρίων που σημαίνει ταχύτατη, βραχυπρόθεσμη και πάρα πολύ πυκνή συναλλαγή, πολύ πυκνό αριθμό συναλλαγών με βάση έναν άλλο θα μου πείτε γιατί πρέπει ο χρηματιστή να χρησιμοποιεί αλγόριθμο, γιατί δεν κάνει μόνο του τι συναλλαγέ τη αγοραπολισία. Είναι πολύ απλό ότι είναι τόσες πολλές οι αγοραπολισίε που μπορεί να ε, εκτελέσει ένας αλγόριθμος που ένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε με την ίδια ταχύτητα να ολοκληρώσει. Όλο λοιπόν το σκεπτικό αυτό έχει να κάνει με πολύ μικρό ποσοστό κέρδους σε κάθε συναλλαγή. Ένα ε, ηλεκτρονικός υπολογιστή με ένα κατάλληλο πρόγραμμα λοιπόν μπορεί να κάνει εκατομμύρια τέτοιων συναλλαγών μικρού κέρδου την ίδια στιγμή. Εδώ βέβαια προκύπτουν πολύ βασικά ζητήματα και ερωτηματικά όπως σε παραδείγματι το κύρος τέτοιων συμβάσεων. Και βέβαια τη αστική ευθύνη σε περίπτωση αγοράς, συμβάσεως αγοράς. Εάν λοιπόν υπάρχει αυτό το παράδειγμα, πρέπει να υποθέσουμε και να δεχθούμε ότι τη σύμβαση τη συνάπτει ο αλγόριθμος. Και ο χρηματιστής μπορεί να μην έχει καμία δυνατότητα ελέγχου του τι πράττει ο αλγόριθμος. Με αυτό λοιπόν το παράδειγμα άρχισε να με απασχολεί το ζήτημα της περίπτωσης ένα ρομπότ να θέλει να προβεί σε σύναψη σύμβασης. Και έτσι πάω στο επόμενο βήμα που είναι η απορία τι απαιτείται για να συναυθεί μία σύμβαση. Χρειάζεται λοιπόν πρόσωπο με νομική προσωπικότητα και, δικαίωμα, και, και ικανό προς δικαιοπραξία που μπορεί να ασκεί τα δικαιώματά του. Αυτές είναι γνωστές έννοιες του δικαίου Βέβαια κύριο μέλημα δικό μου είναι το εξή: ότι για να συναυθεί συμφωνία χρειάζεται η εκδήλωση βούλησης ή η ανταλλαγή ε, προσφοράς και αποδοχή ε, που είναι αντίστοιχη με την εκδήλωση της βούλησης, με τη δήλωση της βούλησης. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε αν το ρομπότ, ο αλγόριθμο, το πρόγραμμα στον ηλεκτρονικό υπολογισμό είναι σε θέση να προβεί σε δήλωση βουλήσεως. Μπορεί φερειπίν το ρομπότ να, να εκδηλώσει πρόθεση για ε, συμμετοχή σε μια συμβατική ε, σχέση. Μπορεί αυτό να ανήκει σε, στον τομέα της ε, επιστημονικής φαντασίας γιατί δεν έχει νομική προσωπικότητα το ρομπότ. Δεν αναγνωρίζεται δηλαδή ως νομικό πρόσωπο από το αστικό δικαίωμα και, και άρα δεν μπορεί να ε, καταστεί συμβαλόμενο μέρος σε μια σύμβαση αυτόνομα. Αλλά αλλάζει το πράγμα εάν κοιτάξουμε διαφορετικά την υπόθεση ενός ρομπότ, αλγορίθμου και το καθεξής το οποίο ε, ε, δηλώνει τη βούληση να προβεί σε σύμβαση εξ ονόματος κάποιου άλλου. Από την ανάπτυξη λοιπόν του σχετικού συστήματος προγραμματισμού μπορούμε να κάνουμε διάκριση μεταξύ του ρομπότ που μπορεί αυτόβουλα να λάβει απόφαση διδασκόμενο από την εμπειρία του και εκείνου που δεν έχει αυτονομία βούλησης. Άρα το κύριο ζήτημα είναι μπορεί ένα ρομπότ ή ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή να ε, δηλώσει βούληση, να προβεί σε δήλωση βουλήσεως, αυτονόμως. Όταν πρόκειται για μη περίπλοκους αλγορίθμους, νομίζω ότι η κατάσταση και η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Όταν χρησιμοποιώ έναν υπολογιστή, Φερρυπίν. Χρησιμοποιώ προγράμματα, τρέχω προγράμματα με μη περίπλοκους αλγορίθμους και θα έλεγα ότι μπορούμε να κάνουμε την εξής ε, ε, παρομοίωση. Ο μη περίπλοκος αλγορίθμος είναι κάτι σαν να γράφω μια επιστολή. Εάν δηλαδή χρησιμοποιώ ηλεκτρονικό πρόγραμμα στον υπολογιστή μου για να απευθύνω μια επιστολή στον πρόεδρο της Επιτροπής, ένα ηλεκτρονικό μήνυμα δηλαδή, θα ήταν σαν να, έγραφα, σαν να έκανα μια χειρόγραφη επιστολή. Απλά τα πράγματα. Είναι πιο περίπλοκα όμως στην περίπτωση του high frequency trading, των ε, ε, συναλλαγών, ε, χρηματιστηριακών συναλλαγών υψηλής συχνότητας, όπου για λόγους νομικούς τα προβλήματα περιπλέκονται και γιατί μπορεί εκεί ένα τέτοιο πρόγραμμα να μην έχει καν αντίληψη του τύπου συμβάσεως την οποία συνάπτει, την ώρα που τη συνάπτει. Άρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για δήλωση βουλήσεως από τον, από χρηματιστή, ο οποίος δεν είχε μπορέσει να προβλέψει πιθανή αγορά ή εν πάση περιπτώσει άλλη σύμβαση ή αντικείμενο συμβάσεως. Πώς μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι έχει προβεί σε μια επαρκή δήλωση βουλήσεως ή προθέσεως. Άρα πρέπει να διερωτηθούμε τι απαιτείται για να είναι πλήρης η βούληση εν ώψη της συνάψεως μιας σύμβασης. Η δήλωση σύμβαση, η ε, βούληση είναι η εξωτερική εκδήλωση της απόφασης για ε, μία ε, συμφωνία η οποία θα έχει νομικές συνέπειες. Δηλαδή η βούλησή μου να καταστώ συμβαλόμενο μέρος σε μία σύμβαση. Εάν λοιπόν έχω ένα περίπλοκο μηχάνημα, ένα ευφιέ e ψυγείο ή έναν αλγόριθμο, που είπαμε νωρίτερα, που μπορεί να αγοράσει και να πουλάει μετοχές. Μπορεί να έχει τη βούληση για σύναψη μια συγκεκριμένη ενοχική σχέση. Να το, να το πω και διαφορετικά. Με το να πατήσω το Enter στο πληκτρολόγιο μου, εγώ ο προγραμματιστής ή για το πρόγραμμα μπορώ να θεωρήσω ότι έχει επαρκή δήλωση βούλησης εκφραστεί είτε ως προσφορά είτε ως αποδοχή με, με όρους αστικού δικαίου. Νομίζω ότι αυτό το ζήτημα δεν έχει ακόμα κρυθεί. Βεβαίω μπορεί κανείς να πει ότι θα πρέπει ο αποδέκτης της δηλώσεως βουλήσεως να είναι εκείνος τον οποίο θα προστατεύσει περισσότερο το δίκαιο, δηλαδή η ιδέα της εμπιστοσύνης στις συναλλαγές, της πίστης, ή μπορεί να ακολουθήσουμε υποκειμενική προσέγγιση. Αλλά για μένα δεν είναι ξεκάθαρο το ποιο μέρος θα είναι αυτό στο οποίο θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη προσοχή στην διαδικασία αυτή της εκδήλωσης μιας βούλησης και αν πρέπει στο χρήστη να δώσουμε περισσότερη, περισσότερο βάρος, παραδείγματι. Ε, ένα άλλο παράδειγμα, με ένα ευφυές ψυγείο το οποίο αποφασίζει ότι θα στείλει μια παραγγελία το οποίο στέλνει μια παραγγελία για ε, αγορά προϊόντων. Ο αντισυμβαλόμενος γνωρίζει, έχει επαρκή γνώση του ποιος είναι εκείνος ο οποίος αποστέλει την σχετική παραγγελία. Είναι επαρκή δηλαδή η έκφραση τη βούληση. Και σε σχέση με τα αυτόνομα ρομπότ. Εδώ έχουμε να κάνουμε με πράξη η οποία δεν εμπλέκει πουθενά δήλωση προθέσεως από πρόσωπο. Αν έχουμε ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικό του υπολογιστή το οποίο έχει να κάνει με τεχνητή νοημοσύνη και το οποίο αφήνει στην ε, ε, επιλογή ενός μηχανήματος την ε, αποστολή μιας παραγγελίας δεν υπάρχει δήλωση βουλήσεως από το πρόσωπο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με συγκεκριμένε δηλώσεις ε, βούλησης όπως απαιτείται από το αστικό δίκαιο. για να υπάρξει ενοχή πρέπει να υπάρχει η εκδήλωση μιας πρόθεσης για ε, σύναψη ενοχικής σχέσης. Βεβαίως θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι έχει συνέπειες νομικές η ένομες συνέπειες, η ε, πράξη αυτού του εφιούς ψυγείου ή ουδήποτε άλλο ρομπότ ή τεχνητού, τεχνικού, τεχνητής νοημοσύνης μηχανήματος, με τη διαφορά όμως ότι αυτά δεν έχουν νομική προσωπικότητα. Και άρα τίθεται ζήτημα αμφισβήτησης του κύρους της συμβάσεως αυτής που έχει συναφθεί χωρίς την βούληση του χρήστη. Και αυτό που θα ήθελα εν τέλει να μείνει από την παρουσίασή μου είναι ότι από τη θεώρηση του αστικού δικαίου, του ενοχικού δικαίου συγκεκριμένα, τα πράγματα περιπλέκονται ιδιαίτερα όταν έχουμε να κάνουμε περιπλέκους αλγορίθμους και προγράμματα. Όταν έχουμε να κάνουμε απλούς αλγορίθμους και προγράμματα είναι απλό και ευχερές να ε, εντοπιστεί η βούληση και η εκδήλωση της βουλήσεως για τη σύναψη μιας σύμβασης. Ε, όταν όμως φτάνουμε σε ένα στάδιο που ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα παίρνει στη θέση μας απόφαση για τη σύναψη μιας σύμβασης που δεν έχει όμως το ηλεκτρονικό αυτό πρόγραμμα ε, νομική προσωπικότητα, δεν μπορεί να ασκήσει κανένα δικαίωμα, τότε υπάρχει ζήτημα σοβαρό κύρους της συμφωνίας. Και επισημαίνω ότι υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις ως προς την ε, αντιμετώπιση των ζητημάτων των συμβάσεων μεταξύ μηχανών machine to machine contract και της ε, αστικής ευθύνης. Αλλά τα πάντα νομίζω θα προκύψουν αφού ξεκαθαρίσει το θέμα των ορισμών. Ήταν για μένα πολύ δύσκολο να προβώ στη διάκριση που θα πρέπει αυτές οι περίπλοκες έννοιες να χρησιμοποιούνται, δηλαδή πού, γίνεται, πού, πού εντοπίζουμε την ε, τεχνητή νοημοσύνη, από πού αρχίζει ο περίπλοκος αλγόριθμος που λαμβάνει εντοπιζουμε αποφάσεις και πού τελειώνει ο απλός αλγόριθμος. Αυτό είναι για μένα το πιο δύσκολο νομίζω, οι ορισμοί και οι διακρίσεις ε, των κατηγοριών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να ακούσουμε και άλλη μια παρουσίαση και συνεχεία να ακούσουμε ερωτήσεις και τις απαντήσεις σε αυτές. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο δόκτωρ Ανδρέα Μπερτολίνη από τη Σκόλα Σουπεριόρε Σαντάνα και το Πανεπιστήμιο της Πίζας. Θα μιλήσει για την ευθύνη και τη διαχείριση του κινδύνου στη ρομποτική. Έχετε το λόγο. Να προβληθεί μου παρακαλώ οι διαφάνειες μου. Να ξεκινήσω. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση καταρχάς. Με χαρά μου ήρθα εδώ. Ως Ευρωπαίος πολίτης χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ασχολείται με αυτό το πολύ επίκαιρο θέμα και συζητάει με ένα πιο συστηματικό τρόπο, πολύ πιο συστηματικό από άλλες μεγάλες οικονομίες. γιατί είναι ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει όλο τον κόσμο και θα υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό στο μέλλον. Λοιπόν, η παρουσίασή μου βασίζεται σε τρεις άξονες. Πρώτον, θα προσπαθήσω να εξηγήσω γιατί πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε μια λειτουργική προσέγγιση στη ρύθμιση των, της ρομποτικής ε, εν συνεχεία θα σας πω ότι τα ρομπότ είναι προϊόντα και προκύπτει το ερώτημα εάν οι τρέχοντες κανόνες, ειδικά για την ευθύνη των προϊόντων που έχουμε στην Ευρώπη, είναι επαρκείς για να διαχειριστούν αυτή την επανάσταση της ρομποτικής. Και τέλος θα μιλήσω για την, το πέρασμα από την ιδέα της αξιολόγησης ευθύνης στη διαχείριση του κινδύνου. Καταρχάς τι είναι τα ρομπότ και πώς πρέπει να τα ορίσουμε. Ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν μπορεί να υπάρχει ένας ορισμός που να τα καλύπτει όλα τα ρομπότ. Είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους ε, μηχανές. Και γιατί ο, ρομπότ, ε, το όρος ρομπότ είναι τεχνικός, ε, προκύπτει δεν είναι τεχνικός μάλλον, προέρχεται από την επιστημονική φαντασία. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν διάφορα είδη, ας πούμε, ε, αυτό το ρομπότ, ας πούμε, το οποίο αυτόνομα οδηγεί ένα αυτοκίνητο, που, αυτό που χρησιμοποιούμε στο χειρουργείο, ε, ένα σύντροφο ρομπότ, ας πούμε, που, που ζει στο καθημερινό μας ε, περιβάλλον, αυτέ αυτές τις εφαρμογές δεν μπορούμε να τις θεωρήσουμε ότι είναι το ίδιο πράγμα. Δεν μπορούμε να τις ρυθμίσουμε με τον ίδιο τρόπο, θα πρέπει να ρυθμίσουμε τα επιμέρους θέματά τους χωριστά. Γιατί οι διαφορές αυτές τις ομάδες εφαρμογών είναι ε, πολύ πιο σημαντικές από τις ομοιότητές τους και άρα θα πρέπει να εστιάσουμε στα προβλήματα που προκύπτουν όταν προσπαθούμε να εφαρμόσουμε τους ισχύοντες κανόνες σε αυτές τις διαφορετικές ε, ομάδες εφαρμογών. Επίσης τα προβλήματα που μοιάζουν παρόμοια, αν δεν είναι ταυτόσιμα, ειδικά το θέμα της ευθύνη, ε, το πιο Ποιο πληρώνει για την ευ... ζημιά όταν κάτι πάει κακά. Μπορεί να πετούν διαφορετικέ τεχνικέ λύσει. Δηλαδή, νομικές εννοώ εδώ, ανάλογα με την ε, εφαρμογή για την οποία μιλάμε. Το ρομπότ για το οποίο μιλάμε. Θα μιλήσω λοιπόν για τους κανόνες ε, ευθύνη. Ποιο πληρώνει δηλαδή για τις ζημιές όταν κάτι δεν πάει καλά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί οι κανόνες για την ε, ευθύνη ε, καθορίζουν ε, και το ποιος πληρώνει αλλά και τι ε, καθορίζουν τελικά και τα κίνητρα που έχουν ε, οι παραγωγοί, ας πούμε, για να αναπτύξουν νέε συσκευέ. Άρα τα κίνητρα που δίνονται στην Ευρώπη, που έχουμε καλή τεχνολογική έρευνα, ε, που χρηματοδοτείται καλά από ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά θα πρέπει αυτά τα προϊόντα, αυτή την καινοτομία, την ε, προχωρήσουμε μέχρι την αγορά, ούτω ώστε να την εκμεταλλευτούμε οικονομικά και κοινωνικά. Θα πρέπει λοιπόν να υιοθετήσουμε καινοτόμε προσεγγίσει στην νομοθεσία. Η καινοτομία να μην, δεν περιορίζεται μόνο στι τεχνολογικέ πτυχέ, είναι και νομική καινοτομία. Και αυτό που θα πρέπει να μα απασχολήσει είναι η εκ των προτέρων βεβαιότητα. Γιατί αν δεν υπάρχει αυτή η βεβαιότητα, οι ερευνητέ και οι παραγωγοί δεν μπορούν να επενδύσουν ε, και να αναπτύξουν αυτέ τι τεχνολογίε ε, και να φτάσουν αυτέ τι τεχνολογίε στην αγορά. Επομένω, κινδυνεύουμε ε, να έχουμε ένα νεφελώδε νομικό σύστημα και να δημιουργήσουμε μία αβεβαιότητα, ούτω ώστε οι καλέ ευρωπαϊκέ ιδέε να μην γίνουν ποτέ καλά ευρωπαϊκά προϊόντα. Επομένω, τα ρομπότ είναι προϊόντα. Πιστεύω ότι δεν πρέπει σήμερα να σκεφτόμαστε ηλεκτρονικές προσωπικότητες και τέτοια. Θα πρέπει ε, να δούμε ποιος άνθρωπος θα είναι ο υπεύθυνος για την ε, ζημιά που κάνει η μηχανή. Και θα είναι είτε ο χρήστης είτε ο ιδιοκτήτης, που μπορεί να είναι και διαφορετικοί αυτοί οι δύο, αλλά μπορούμε να τους βάλουμε μαζί ας πούμε, στην ομάδα, ή ο παραγωγός, δηλαδή αυτός που έχει λόγο για το πώς αναπτύσσεται το προϊόν, τι χαρακτηριστικά έχει κτλ. Εάν τα ρομπότ προϊόντα, οι κανόνες για την ευθύνη των προϊόντων ισχύουν και ιδίω η οδηγία ε, του 85, 374 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα, ε, υπάρχει αρκετά χρόνια τώρα, αλλά δεν έχει καλή επίπτωση ε, στην ευρωπαϊκή αγορά και θα σας εξηγήσω πολύ γρήγορα γιατί. Ο παραγωγής θεωρείται υπεύθυνο όταν υπάρχει πρόβλημα παραγωγής, ένα πρόβλημα με την προειδοποίηση ή ένα ε, ελάττωμα ας πούμε, στο σχεδιασμό που δημιουργεί βλάβη σε κάποιον. Ε, αυτό έχει να κάνει με την καινοτομία. Γιατί, δηλαδή, α, λέμε, είναι σαν να λέμε ότι αν το προϊόν ε, είχε σχεδιαστεί διαφορετικά θα ήταν πιο ασφαλές. Τώρα, ε, ο σκοπός των κανόνων ε, ευθύνης είναι διτός. Καταρχάς να δώσουμε κίνητρα τους ώστε να είναι ασφαλές το σχέδιο. Θέλουμε οι παραγωγή να φτιάχνουν προϊόντα καλής ποιότητας και ασφαλή τους Ευρωπαίους χρήστες και θέλουμε επίσης ε, να διευκολύνουμε το θύμα, να του δώσουμε δηλαδή άμεσα αποζημίωση. Αυτή είναι η... Από τη μία έχουμε λοιπόν την αυστηρή ευθύνη ή την απλή αμέλεια από την άλλη ας πούμε. Ε, ε, θα πρέπει να υπάρχει σχέση του ανάμεσα στην ζημία, ας πούμε, και στο ελάττωμα και να αποδειχθεί, ας πούμε, τόσο ο παραγωγός να είναι υπεύθυνο. Όμως υπάρχουν κάποια προκαταρτικά στοιχεία τα οποία ε, ερευνώ και που δείχνουν ότι αυτοί οι κανόνες δεν λειτουργούν πολύ καλά. Καταρχάς, αυτοί οι κανόνες που έχουμε εδώ στην Ευρώπη ε, μοιάζουν με αυτούς τους, ε, Αμερικής, αλλά έχουν τελείως διαφορετικά, έχουμε τελείως διαφορετικά επίπεδα νομικών διαφορών εδώ και στην Αμερική. Δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε ε, λέγοντας ότι τα δικά μας προϊόντα είναι πολύ πιο ασφαλή από τα αμερικάνικα, γιατί στην πραγματικότητα είναι περίπου τα ίδια. Ο λόγος έχει να κάνει προφανώς με το νομικό μας σύστημα, το δικό μας και των Αμερικανών. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στην ευθύνη με βάση το, τους κανόνες για την ε, ε, ευθύνη των προϊόντων ή την ασφάλεια πούμε, των προϊόντων κτλ. Ε, οι ενάγοντες στην Ευρώπη ε, σπάνια ε, έχουν επιτυχία, ας πούμε. Άρα οι κανόνες στην Ευρώπη δεν είναι επαρκείς για να προστατεύσουν τον καταναλωτή. Γιατί ε, οι νομικές διαφορές, οι δίκες κτλ. είναι περίπλοκες και ε, πολύ ακριβές, πούμε. Ε, είναι δύσκολο να αποδείξει, ας πούμε, τη σχέση του, δηλαδή τη, τη ζημιά του που υφίστασε και την ευθύνη, α πούμε. Είναι πρόβλημα για τη ρομποτική. Προφανώ. ειδικά για τη ρομποτική. Γιατί οι κανόνε στη ρομποτική ε, μετατοπίζουν ε, την ευθύνη από τον ε, χρήστη και τον ιδιοκτήτη στον παραγωγό. Και αυτή η, μεταβίβαση οφείλεται στον αυτοματισμό. Αν, ας πούμε, ένα όχημα δεν έχει οδηγό. Σήμερα, ας πούμε, ο οδηγός θεωρείται ε, υπεύθυνο. Αλλά όσο πιο αυτόματη είναι η διαδικασία οδήγησης, τόσο πιο πολύ θα φταίει ο παραγωγός. Αυτή η μετάβαση όμως δεν θα γίνει εν μία νυχτή. Θα υπάρξει μια μακρά βάση όπου δύο διαφορετικοί κανόνες, δηλαδή ε, αυτοί που θα θεωρούν τον ε, ε, χρήστη και αυτοί που θα θεωρούν τον παραγωγό υπεύθυνο, θα αλληλεπικαλύπτονται και θα δημιουργούν και αβεβαιότητα και περίπλοκες νομικέ διαφορέ, Γι' αυτό φοβούνται εδώ, αυτό φοβούνται οι παραγωγοί και οι ασφαλιστικέ εταιρείε. Ε, γιατί θα είναι δύσκολο να προσωπικοποιήσουμε ας πούμε, τον ε, κίνδυνο που υφίσταται ένας ε, χρήστης και επομένως τι, τι, τι πρέπει να καλύπτουν οι ασφαλιστικέ εταιρείε. Αυτό σημαίνει καθυστέρηση για την καινοτομία, δεν θα φτάσουν γρήγορα τα προϊόντα στην αγορά, τα καινοτόμα κτλ. Και ένα δεύτερο φαινόμενο πρέπει να λάβουμε υπόψη. Χάρη στην αυτοματοποίηση και στην ανάπτυξη τη τεχνολογία τη. Σα παρακαλούμε λίγο πιο αργά. Υπάρχει μια μετάβαση προς τους κανόνες ε, ευθύνη των προϊόντων σε τομείς που σήμερα ρυθμίζονται μέσω άλλων κανόνων. Φερρυπίνη. Ας πούμε το ιατρικό λάθος. Σήμερα υπάρχουν απίστευτες ε, νομικές διαφορές ε, κατά των γιατρών, ας πούμε, δίκες κατά των γιατρών, όταν ας πούμε δεν θεραπεύουν σωστά έναν ασθενή. Εάν βάλεις τώρα και την τεχνητή νοημοσύνη στο σύστημα απόφασης, και, θα, υπάρχει αυτή η τεχνολογία, το ξέρουμε, ε, τότε θα έχουμε μια μετάβαση. Μερικές φορές ο παραγωγός ας πούμε, του τεχνητού συστήματος, ε, της τεχνητής νοημοσύνης ας πούμε, ε, είναι υπεύθυνο ε, ή ο, άλλες φορές ο γιατρός. Ας πούμε το ίδιο και στα τροχέα. Αυτή τη αυξηθεί η αυτοματοποίηση στην οδήγηση, τότε θα σταματάμε να μηνύουμε ας πούμε τον οδηγό ε, και θα μηνύουμε την εταιρεία. Εάν οι κανόνε για την ευθύνη των προϊόντων δεν λειτουργούν όπω πρέπει, τότε θα δημιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την ανάπτυξη ε, τη ρομποτική στην Ευρώπη. Ε, Επομένω, τι προτείνω για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα πολύ περίπλοκα θέματα. Εγώ προτείνω να ξεκινήσουμε τα εξή να κάνουμε τα εξή πράγματα. Καταρχάς, η ασφάλεια είναι καλύτερη ε, μέσω της εκ των προτέρων τυποποίηση. Πιστεύω ότι οι κανόνε ευθύνε δεν είναι πολύ αποτελεσματικά για να εξασφαλίσουν τα προϊόντα τα οποία πολλούνται στην ευρωπαϊκή αγορά είναι ασφαλή. Νομίζω ότι αν είχαμε καλύτερα ε, τεχνολογική τυποποίηση θα είχαμε καλύτερο αποτέλεσμα. Παράλληλα, δεν θα πρέπει να μας απασχολεί τόσο πολύ το να ε, ρίξουμε το φταίξιμο σε κάποιον που έκανε κάτι λάθος. Αυτό είναι το παραδοσιακό κόνσεπτ της ευθύνη. Θα πρέπει να έχουμε διαφορετική προσέγγιση. Δηλαδή από την οικονομία να εμπνευστούμε και να δώσουμε την ευθύνη στο μέρος το οποίο βρίσκεται πολύ πιο κοντά σε καλύτερη θέση για να μειώσει το κόστος και μέσω της ασφάλισης. Και επίσης θα πρέπει να έχουμε ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις δοκιμές στο ρομπότ. Λοιπόν, τεχνολογική τυποποίηση καταρχάς. Θα πρέπει να έχουμε ε, ευρωπαϊκά τεχνικά πρότυπα για τα ρομπότ. Όλες τις μεγάλες οικονομίες θα πρέπει ε, γρήγορα να αναπτύξουν τα δικά τους τεχνολογικά πρότυπα και να τα ανεβάσουν. Ε, αν το κάνουμε πρώτοι θα έχουμε μια ε, κυρίαρχη θέση στην αγορά. Χρειαζόμαστε να ενισχύσουμε τέλο πάντων αυτό το ευρωπαϊκό επίπεδο τεχνολογικής τυποποίησης. Και για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να αναπτύξουμε ε, τεχνολογικά πρότυπα πολύ συγκεκριμένα που θα επικροτηποιούνται πολύ συχνά και που θα είναι πολύ συγκεκριμένα για διαφορετικές εφαρμογές. Για να το κάνουμε αυτό μπορούμε να ε, έχουμε, έχουμε, έχουμε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Τυποποίησης αλλά μπορούμε να αναδαθμίσουμε το ρόλο της ή αλλιώς μπορούμε να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ρομποτικής με ακριβώς αυτό το καθήκον, να αναπτύξει δηλαδή τεχνολογικά πρότυπα τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη και δοντολογικές πτυχές, ηθικές πτυχές, που είναι σημαντικές. Αλλά σήμερα αν μιλήσεις, για, μιλήσεις με μηχανικούς θα σου πούν ότι δεν έχουν σαφώς τεχνολογικά πρότυπα που να ξέρουν πώς, ε, που να τους καθοδηγούν για να αναπτύξουν κατάλληλα προϊόντα. Ε, αν δεν το κάνουμε εμεί, το κάνει κάποια άλλη μεγάλη οικονομία, οι Αμερικανοί ή κάποιοι άλλοι. Και αυτή τη στιγμή ε, υπάρχουν αυτά τα πρότυπα, θα τα υιοθετήσει ο κλάδο. Αν τα υιοθετήσουμε εμεί, λοιπόν, θα είμαστε σε καλύτερη θέση. Το να έχει την ευθύνη το μέρο το οποίο ε, είναι σε καλύτερη θέση για να μειώσει το κόστο. Το χειρότερο ποιο είναι η αβεβαιότητα, γιατί από την αβεβαιότητα προκύπτουν διαφορέ νομικέ, ε, δίκε κτλ. Ε, και πολύ δύσκολα θα μπορούν οι ασφαλιστικές εταιρείες να καλύπτουν το, και το κόστος αλλά και να υπάρχουν νέα προϊόντα στην αγορά. Επομένως, θα πρέπει να περάσουμε στην απόλυτη ε, ευθύνη που είναι κάτι παραπάνω από την αυστηρή ευθύνη. Δηλαδή χωρίς τη δυνατότητα ε, να αποδεσμευτείς από αυτήν ε, χωρίς υπεράσπιση ας πούμε. Ε, αυτό φαίνεται, είτε, αν αυτό φαίνεται υπερβολικό βάρος για το χρήστη ή για τον παραγωγό, ανάλογα με την εφαρμογή ας πούμε μπορούμε να δώσουμε διαφορετικές απαντήσεις. Μέσω της, των υποχρεωτικών συστημάτων ασφάλισης επίσης μπορούμε να διαχειριστούμε το κόστος αυτό. Και θα μειωθεί συνολικά το κόστος, δεν θα αυξηθεί το κόστος. Και επίσης, αν είναι σαφές αν α πούμε έχουμε έναν κατασκευαστή αυτοκινήτου όπου θεωρείται 100% για όλες τις ζημιές που απορρέουν από τη χρήση του οχήματό του, μπορεί να ασφαλίσει αυτόν τον κίνδυνο σε μια ασφαλιστική εταιρεία και μπορεί αυτό το κόστος να το ενσωματώσει στο κόστος παραγωγής και να το, διανύμει αυτό, το, να το κατανείμει αυτό το κόστος μεταξύ όλων των χρηστών της τεχνολογίας μέσω μηχανισμών ε, τιμών κατά τη στιγμή πώληση των αυτοκινήτων του. Και τέλος, Χρειαζόμαστε ένα νέο πλαίσιο για τις δοκιμές των ρομπότ σε πραγματικά ε, αληθινά σενάρια. Είμαστε πολύ καθυστερημένοι. Στην Ιαπωνία έχουν, ας πούμε, εδώ και αρκετά χρόνια τις ε, λεγόμενες ειδικέ ζώνες τόκου όπου ε, επιτρέπονται οι δοκιμές ρομπότ σε σενάρια που συναντάμε ας πούμε στην πραγματική ζωή. Πρέπει να δοκιμάσουμε, πρέπει να τεστάρουμε τα ρομπότ ε, εκτός των εργαστηρίων για να δούμε πώς θα αντιδράσουν όταν αλληλεπιδρούν με τα ανθρώπινα όντα. Είναι πάρα πολύ περίπλοκο αυτό όταν κάποιο προσπαθεί να καινοτομήσει, γιατί οι κανονισμοί σε όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε ε, δεν είναι οι ίδιοι και δεν υπάρχουν σαφεί κανόνε που να λένε πότε και υπό ποιε συνθήκε ε, θα πρέπει να γίνεται μια δοκιμή, να επιτρέπεται μια δοκιμή. Το κάνουν όμω στην Ιαπωνία, το κάνουν στι ΗΠΑ και επομένω θα πρέπει να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε κι εμεί. Και νομίζω ότι καλό θα ήταν να υπάρχει μια νομοθεσία εδώ πέρα θα βελτίωνε συνολικά τη θέση της ε, ευρωπαϊκής ε, βιομηχανίας, ειδικά αυτή που προσπαθεί να καινοτομήσει. Θα μας βοηθούσε να εντοπίσουμε και τους ε, κινδύνους που θα μπορούσαμε να τους διαχειριστούμε μέσω ασφάλισης και μέσω καλύτερων κανόνων ευθύνη, ούτω ώστε να περάσουμε από την έρευνα για τη ρομποτική στην Ευρώπη στην κατασκευή ρομποτικών μηχανημάτων. Ευχαριστώ πολύ για τις πολύ ενδιαφέρουσες θέσεις σας. Ως Τσέχος πιστεύω ότι αυτός ο οργανισμός ε, ρομποτικής θα έχει την έδρα του στην Πράγα, γιατί ξέρετε ότι η λέξη ρομπότ είναι τσεχική, που σημαίνει εργάτης. Και όπως είδαμε υπάρχει η πιθανότητα να καταλήξουμε και σε κάτι τέτοιο ρομπότ εργάτης δηλαδή. Η κυρία Ντελβό έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για την ε, παρουσίαση και για τις δύο παρουσιάσεις. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Έχω ένα ερώτημα για την ευθύνη. Είπατε ότι θα, θα, θα βαρύνει είτε τον χρήστη είτε τον κατασκευαστή. Αλλά Βλέπω ότι υπάρχουν και διάφοροι ενδιάμεσοι. Ένα αυτόνομο αυτοκίνητο, για παράδειγμα, χρειάζεται πληροφορίες οι οποίες του παρέχονται μέσω αισθητήρων. Τι συμβαίνει αν, για παράδειγμα, δεν καταφτάσουν έγκαιρα οι πληροφορίες στο αυτοκίνητο, στον εγκέφαλο του αυτοκίνητου. Ποιος βαρύνεται με την ευθύνη σε αυτή την περίπτωση. Ε, όταν δηλαδή υπάρχουν ενδιάμεση μεταξύ του κατασκευαστή και του τελικού χρήστη. Και μετά έχω και ένα ερώτημα για τους αλγόριθμους. Οι αλγόριθμοι ε, συνήθως ε, είναι απλοί στην κατανόηση για τους απλούς ανθρώπους, για τους κανονικούς ανθρώπους. Άρα τι, τι, τι ισχύει σε σχέση με τη διαφάνεια γύρω από αυτούς τους αλγόριθμους. Υπάρχουν ζητήματα που σχετίζονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, για παράδειγμα. Αυτά είναι τα δύο ερωτήματα που έχω. Και πρέπει να σας πω ότι πραγματικά βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα την παρουσίασή σας. Θα, λέω, Πρόεδρος, θα πάρουμε πρώτα τις ερωτήσεις και στη συνέχεια θα σας δώσω το λόγο να απαντήσετε. Κύριε Κομοντίνη, ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους προσκεκλημένους μας για τις εξαιρετικές παρουσιάσεις τους που μας εμπνέουν όπως είπε και η κυρία Ντελβό. Έχω δύο ερωτήματα που σχετίζονται ε, ένα για τον ε, κύριο από τη Βαρσοβία που σχετίζεται με την ευθύνη, ε, την αστική ευθύνη και τους αλγόριθμους. Πρώτον, αν ο χρήστης χρησιμοποιεί αλγόριθμο, όπως για παράδειγμα ε, ο χρηματιστής. Η ευθύνη δεν είναι παρόμοια με την έννοια αστικού ε, δικαίου ότι ο χρηματιστής ε, είναι εκείνος που βαρύνεται με την ευθύνη σε περίπτωση ζημίας. Και δεύτερον, αν υπάρχει αυτόνομο ρομπότ και του δώσουμε και ηλεκτρονική προσωπικότητα νομικής φύσεως, αυτό μπορεί να τελικά να εκδηλώνει βούληση σε νομικές συναλλαγές, να να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε να απευθύνετε ερωτήματα και στον κύριο Κρατικόφσκι. Να πω πρώτα για το ζήτημα του, των ενδιαμέσων. Το πρώτο που πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι θέλουμε να δίνεται αποζημίωση στο θύμα. Γιατί το θύμα σίγουρα δεν ευθύνεται. Ε, και έτσι ε, δικαιούται αποζημίωση. Άρα πρώτος στόχος είναι να δίνεται αποζημίωση στο θύμα. Για να γίνει αυτό θα θεωρούσα ότι θα πρέπει να θεωρείται υπεύθυνο ο ε, κατασκευαστής. Ακόμη και αν ευθύνεται κάποια, κάποιο στοιχείο ή κάποια πληροφορία που παρεσχέθη από τρίτον αυτό σχετίζεται με την διαχείριση ε, κινδύνου. Γιατί αν ευθύνεται στο 100% των περιπτώσεων ο κατασκευαστής, αυτός θα πρέπει να αποζημιώνει το θύμα που πραγματικά δεν φέρει καμία ευθύνη. Ταυτόχρονα, ο κατασκευαστής μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας ε, και του, του ασφαλιστηρίου συμβολέου του και τις συμβατικές ε, του υπηρεσίες που παρέχει, θα μπορούσε να συνάψει συμβατικές σχέσεις βάσει των οποίων θα μπορούσε να μεταφέρει αυτό το κόστος ε, στον ενδιάμεσο. Διαφορετικά θα δημιουργήσουμε ένα εξαιρετικά περίπλοκο σύστημα όπου ένας μεμονωμένος χρήστης που ε, ε γίνεται θύμα θα πρέπει να προσφεύγει και κατά του κατασκευαστή και κατά όλων των ε, ενδιαμέσων και των προμηθευτών του κατασκευαστή. Θα βρεθεί δηλαδή σε μια πάρα πολύ περίπλοκη κατάσταση από άποψη προσφυγής ε, και ε, είναι λογικό ότι ενδεχομένω να μην έχει ούτε τα κίνητρα ούτε και τα μέσα για να κάνει όλε αυτέ τι προσφυγέ. Οπότε θα βρεθεί σε δινή θέση. Αντιθέτω, αν ο κατασκευαστή ευθύνεται στο 100% των ε, περιπτώσεων και πούμε δηλαδή ότι ό,τι και αν γίνει με τα προϊόντα του εσύ φταίει, εσύ ευθύνεσαι, τότε θα συνάπτει ασφαλιστήρια συμβόλαια και αυτά θα, θα είναι τμήμα όλων των συναλλαγών που κάνει και με τους δικούς του προμηθευτές, δηλαδή τους ε, ενδιαμέσους. Άρα, ε, πρέπει να πούμε ότι όσο πιο, δι... όσο πιο προηγμένες ε, και περίπλοκες γίνονται αυτές οι μηχανές, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να καθορίζεται ποιος ακριβώς ευθύνεται για την πληροφορία που χάθηκε κτλ. Οπότε ε, είναι ενδιαφέρον να, ε, να πούμε ε, ότι το σημαντικό είναι να δίνεται άμεσα η αποζημίωση και το κόστος που προκύπτει να ε, ρυθμίζεται μέσω συστημάτων ασφάλισης. Γιατί με τις προσφυγές που θα μειώσουμε, θα μειώσουμε και το κόστος. Και έτσι θα έχουμε ένα σύστημα πολύ πιο σαφές, πολύ πιο εύχριστο για τους Ευρωπαίους καταναλωτές, αλλά και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Καταρχάς θα ήθελα να δώσω απάντηση στην πρώτη ερώτηση της διαφάνειας στην χρήση των, κατά την χρήση των αλγορίθμων. Και δεν το έχω πει μέχρι τώρα, αλλά είναι πολύ σημαντικό θέμα νομίζω και για μένα. Έχει δικαίωμα και ο χρήστης ασφαλώς να γνωρίζει ότι υπησέρχεται σε μια σύναψη συμβάσεως με αλγόριθμο, αλλά και η άλλη πλευρά έχει δικαίωμα να το γνωρίζει. Και ιδιαιτέρως πιστεύω ότι εάν η κατάσταση φτάσει σε σημείο που θα πρέπει να συζητούμε ε, επαφή με τεχνητή νοημοσύνη, θα χρειαστεί ένα σύστημα καταχώρησης που θα επιτρέπει πρώτα να εντοπίσουμε ε, ότι έχουμε να κάνουμε όχι με άνθρωπο αλλά με πρόγραμμα και να αναγνωρίζουμε ένομες συνέπειες, χαρακτηριστικά δηλαδή αντίστοιχα με αυτά ενός ανθρώπου ή νομική προσωπικότητα στο πρόγραμμα. Για να δώσω απάντηση στη δεύτερη ερώτηση. Αν είναι ανεύθυνο στην επιλογή του προγράμματος ο χρήστη, δεν μπορεί να έχει και την αστική ευθύνη από τις συνέπειε ζημίας που ενδεχομένω έχει προξενήσει αυτό. Ναι, αυτά ως προς την αδικοπραξία. Αυτό όμω, το οποίο, εγώ ανέφερα είχαν να κάνουν με την σύναψη συμβάσεως. Στην περίπτωση λοιπόν ως πολύ περίπλοκου αλγορίθμου έχουμε πραγματική δήλωση βούλησης. Και για να απαντήσω πολύ απλά, χωρίς σχηματισμό ενοχικής σχέσης δεν μπορεί να υπάρξει ούτε αδικοπραξία για μένα. Γιατί νομίζω ότι πήγαμε πολύ μακριά, ε, σε ένα προθύστερο θα έλεγα σχέση με το, με το ενοχικό, γιατί μιλούμε για αδικοπραξία, να πρέπει πρώτα να μιλούμε για ε, ενοχική σχέση. Στην περίπτωση δε που ένας χρηματιστής χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά προγράμματα για τις συναλλαγές του σε μετοχές, μπορεί να έχει αυτός ευθύνη και για ζημία πιθανή. Ε, η απάντηση θα είναι ναι, θα πρέπει να είναι. Ε, θα πρέπει να έχει αστική ευθύνη. Εάν όμως δεν υπάρχει η βούληση, αν δεν μπορεί να εντοπιστεί η βούληση για ενοχική σχέση, πώς μπορούμε να αποδώσουμε αστική ευθύνη στον τομέα του αστικού δικαίου. Γιατί βεβαίως υπάρχει και η άλλη, η άλλη ιδέα της αδικοπραξίας, που είναι ένα άλλο κεφάλαιο και εξήγησε ο συνάδελφος. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Άντερσον έχει ρώτηση. Ναι, για τον δόκτωρα Μπατολίνη. Η πρόταση για την ε, ασφάλιση αυτή ε, έχει ελκυστικά χαρακτηριστικά νομίζω. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες ιδέες πού έχουν ε, ισχύσει αντίστοιχες λύσεις και τι συνέπειες από από αυτές. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, η ασφάλιση είναι ένα ισχυρότατο εργαλείο. Το μόνο θέμα είναι ότι θα πρέπει να καταστεί εξάντε εκ των προτέρων σαφές ποιος και σε ποιο βαθμό μπορεί να θεωρηθεί ε, υπεύθυνο σε αποζημίωση και μέχρι ποιο βαθμό μπορεί να προκύψουν συνέπειες, πρέπει να ποσοτικοποιηθούν οι συνέπειες. Στις οδικές μεταφορές, σε παραδείγμα, έχουν τα περισσότερα κράτη-μέλη εισαγάγει υποχρεωτικό όρο ασφάλισης, που λέει ότι όταν κάποιος αγοράζει αυτοκίνητο θα πρέπει και να ε, αγοράζει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο προκειμένου να καλύπτει ενδεχόμενες ζημίες που έχει, που έχει προκαλέσει το αυτοκίνητό του. Και μάλιστα στην Ιταλία συγκεκριμένα την υποχρέωση αυτή φέρει όχι ο οδηγός αλλά ο ιδιοκτήτης του αυτοκίνητου. Δηλαδή ασφαλίζεται ακόμα και σε ζημία, σε που έχει προκληθεί ανεξάρτητος τη βουλησή του. με τα παραδοσιακά αυτοκίνητα. Σήμερα ξέρουμε ότι όταν προκύψει ένα τρακάρισμα θα φταίει ή ο ένας οδηγός ή ο άλλος. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για υπετιότητα ανθρώπου, ανθρώπινο όντως. Και μπορούμε να προβλέψουμε τι είδου συμπεριφορά μπορεί να οδηγήσει στο ατύχημα, ε, μπορεί να είναι επικίνδυνη οδήγηση, μπορεί να διαγραφεί κάποιο σε μέσα την ώρα που οδηγούσε και ούτω καθεξής. Άρα μπορούμε να τυποποιήσουμε τις συμπεριφορές αυτές, μπορούμε να τις ε, υπολογίσουμε, να τις κατηγοριοποιήσουμε και να τους δώσουμε και μια αξία. Αυτά για χρήση της ασφαλιστικής. Δηλαδή ένας νέος 25 ετών που κατοικεί στην τέτοια περιοχή κτλ. μπορεί να έχει πιθανολόγηση τόση ενώ μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Για τα ρομπότ δεν μπορούμε να το έχουμε αυτό γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε δοκιμή στα ρομπότ σε συνθήκες πραγματικής, πραγματικές, πραγματικής ζωής δεν υπάρχει δυνατότητα για κάτι τέτοιο, τους άλλους δεν υπάρχουν τόσο πολλά ρομπότ. Και, αλλά, αλλά άπαξ και έχουμε αυτά τα δεδομένα, τη συμπίληση των δεδομένων, θα υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος θα μπορεί να ορίσει ένα σαφή κανόνα περί ευθύνης που θα θεωρεί τη μία πλευρά υπεύθυνη κατά 100% ή σε κάποιο ποσοστό και αυτό θα διευκολύνει πάρα πολύ τον χρήστη ε, του ε, αυτοματοποιημένου αυτού μηχανήματος, του ρομπότ. Το πρόβλημα όμως υπάρχει εκεί όπου δεν θα είναι επαρκώς συμφέρουσα οικονομικά η σύναψη μιας, ενός ασφαλιστηρίου συμβολέου για την εταιρεία. Στην προσθετική ρομποτική, παραδείγματι, εδώ έχουμε να κάνουμε μέχρι στιγμή με μηχανήματα τα οποία δεν ξεπερνούν τα, τις ανθρώπινες δυνατότητες. Άρα κάποιος που θα βάλει ένα ρομποτικό πόδι, ένα ρομποτικό χέρι, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν προς το παρόν μία αναπηρία δηλαδή είναι περιορισμένο ακόμα το πεδίο εφαρμογής αυτών των εφαρμογών, των ε, ρομποτικών ε, προϊόντων. Είναι περιορισμένο ο αριθμός των ενδιαφερομένων, ο αριθμός των προϊόντων που θα διατεθούν στην αγορά θα είναι περιορισμένος, η τιμή θα είναι πολύ υψηλή και κατά πάσα πιθανότητα οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν θα ενδιαφέρονται να μπουν στην αγορά. Εκτός και αν τους δοθεί βέβαια κάποιο άλλο είδος, είδους κίνητρο. Θα μπορούσαμε νομοτεχνικά να βρούμε κάποιες άλλες λύσεις βέβαια εφόσον δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη. Ένα ποσοστό παραδείγματι της ε, τιμής του μηχανήματος θα μπορούσε να εισραίει σε ένα διοικητικά οργανωμένο ταμείο το οποίο στη συνέχεια θα χρησιμοποιούνταν για την αποζημίωση των πιθανών θυμάτων της, ε, της λειτουργίας. Άρα δεν θα, θα αποφεύγαμε τη λεγόμενη αποτυχία της αγοράς, το market failure, όπου δεν θα δραστηριοποιηθούν οι ασφαλιστικές εταιρείες γιατί δεν θα έχουν τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση όπως σας είπα και προς το παρόν μόνο θεωρητικά συμφέρον. Και άρα τότε μπορεί να μην αρκούν οι κανόνες του ασφαλιστικού δικαίου και θα ήταν καλό να αναστηθούν άλλες εναλλακτικές υποχρεωτικά ασφαλιστικά συστήματα, παραδείγματι, με σαφή ευθύνη παραγωγού, θα μπορούσαν να καλύψουν ζητήματα που θα προέκυπταν από τα αυτοκίνητα που διαθέτουν αυτόνομη οδήγηση και έτσι και θα βελτιώνονταν τεχνολογικά η αγορά ή το προϊόν. Ευχαριστώ. Καθηγητής με τώρα. Από το... από το Πανεπιστήμιο του Κότεμπορκ θα μιλήσετε για τη ρομποτική, τεχνητή νομοσύνη και τη διαχείριση κινδύνου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου απευθύνατε. Μεγάλη μου χαρά και τιμή που βρίσκομαι εδώ. Η οπτική ε, γωνία από την οποία θα παρουσιάσω εγώ το θέμα μου θα είναι πιο μακροπρόθεσμο. Ίσως κάποιοι ε, θα το θεωρήσετε επιστημονική φαντασία, αλλά σας καλώ να αντισταθείτε σε αυτόν τον πειρασμό, γιατί υπάρχουν ζητήματα που είναι κρίσιμης σημασίας για το κοινό μας μέλλον. Λοιπόν, εδώ μιλώ για την τεχνητή νομοθεσία, για την τεχνητή νοημοσύνη και οι εξελίξεις ε, σε ε, αυτόν τον τομέα θα επηρεάσουν σημαντικότατα την οικονομία. Η έκθεση με McKinsey ε, μάλιστα ε, προέβλεψε ότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρξουν 53 εκατομμύρια δολάρια ωφέλη ε, λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Μακροπρόθεσμα λοιπόν, οι δυνατότητες για την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να φέρουν ευμερία και οι πιθανότητες αυτές είναι απεριόριστες. Ωστόσο υπάρχουν και διάφοροι κίνδυνοι οι τρεις ε, παρακάτω κίνδυνοι θεωρώ ότι είναι οι σημαντικότεροι. Πρώτον, ε, στρατιωτική τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσαν ενδεχομένω ε, τα αεροσκάφη να καταστούν επικίνδυνα αν πέσουν στα χέρια τρομοκρατών. Αυτό είναι η πιο άμεση ενδεχομένως ανησυχία. Δεν αφορά τον, το απότερο μέλλον μετά από δεκαετίες για παράδειγμα. Δεύτερο, robot sourcing. Θα μας εκτοπίσουν τα ρομπότ από την αγορά εργασίας. Και τρίτη ανησυχία, κίνδυνος είναι τι θα συμβεί όταν η τεχνητή νοημοσύνη φτάσει σε ένα επίπεδο όπου εμείς οι άνθρωποι δεν θα είμαστε πλέον τα πιο νοήμονα όντα στον ε, πλανήτη. Θα μπορούσαμε να περιμένουμε ότι θα διατηρήσουμε τον έλεγχο. Εγώ θα μιλήσω για το πιο σημαντικό ε, και το πιο ενδιαφέρον για μένα θέμα, το τρίτο. σχετίζεται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Το ερώτημα λοιπόν είναι, όταν φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη σε αυτό το επίπεδο που εμείς οι άνθρωποι δεν θα είμαστε πλέον τα πιο ευφυή όντα στην γη, θα, έχουμε, θα μπορούσαμε να περιμένουμε ότι θα διατηρήσουμε τον έλεγχο. Σύντομη απάντηση, όχι. Και ε, η συνέπεια είναι ότι η μοίρα μας σε αυτή την περίπτωση και σε αυτό το σημείο θα εξαρτάται από τις προθέσεις των μηχανών. Γι' αυτό θα πρέπει εκ των προτέρων να εξασφαλίσουμε ότι οι προθέσεις αυτών των μηχανών θα, είναι, θα με αυτά που θεωρούμε εμείς σημαντικά, όπως είναι η ανθρώπινη ευημερία για παράδειγμα. Θα ήθελα να περιγράψω τρία επίπεδα ε, καταστροφής. Το πρώτο επίπεδο είναι για παράδειγμα η πυρκαγιά σε ένα σπίτι που μπορεί να είναι τραγωδία σε ατομικό επίπεδο αλλά είναι κάτι που η κοινωνία μπορεί να το χειρίζεται μέσω εταιριών, ασφαλιστηρίων, συμβολέων κτλ. κτλ. Δεύτερο επίπεδο, μεγαλύτερης κλίμακας καταστροφές όπου δεν μπορεί κανείς να περιμένει ότι μία ασφαλιστική εταιρεία θα καλύψει το κόστος. Παράδειγμα εδώ είναι το τσουνάμι και η καταστροφή στο πυρηνικό εργοστάσιο της Φουκουσίμα στην Ιαπωνία. Εδώ χρειάζεται κρατική παρέμβαση, βεβαίως για να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους καταστροφές. Τρίτο επίπεδο ε, έχει μια διάσταση αποκάλυψης. Ε, ποιος θα πληρώσει την ζημιά. Ε, το, τότε, σε αυτή την περίπτωση αυτά τα ερωτήματα δεν μας απασχολούν πια γιατί δεν θα υπάρχουμε εμείς ως άνθρωποι αν γίνει αυτό. Ε, αυτό που συζητούμε σήμερα είναι πώς θα μπορούσαμε να, δια, διασφαλίσουμε ότι δεν θα γίνουν. Δεν θα γίνουν, δεν θα γίνουν τέτοιου είδους πράγματα γιατί από εκεί και πέρα δεν θα, δεν θα χρειάζεται καν να συζητάμε τίποτα άλλο δεν θα υπάρχουμε. Λοιπόν, ε, κορυφαίοι παγκοσμίω επιστήμονες, ε, συμπεριλαμβανομένου του Στέφεν Χόκινγκ, είχαν δηλώσει στον Independent πριν από κανένα δύο χρόνια ότι παρότι οι επιπτώσει τη τεχνητής νοημοσύνης εξαρτώνται από το ποιος την ε, ελέγχει, οι, οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις εξαρτώνται από το αν θα μπορεί γενικά να ελεγχθεί η τεχνητή νοημοσύνη και μπορεί να είναι θελκτικό να απορρίψει κανείς αυτή την ιδέα ως ε, επιστημονική φαντασία, αλλά αυτό ε, θα ήταν σφάλμα να το κάνουμε και ενδεχομένως θα ήταν και το σημαντικότερο σφάλμα της ανθρωπότητας στην ιστορία της. Άρα, ε, η ανθρωπότητα πραγματικά κινδυνεύει, ότι, ε, ε, κινδυνεύει να εξοντωθεί από μηχανήματα. Εξαρτάται από δύο ερωτήματα αυτό. Θα ξεπεραστεί ποτέ η, ανθρώπινη νοημοσύνη από την τεχνητή νοημοσύνη. Και δεύτερον, τι θα τίνουν να κάνουν αυτά τα μηχανήματα τεχνητής νοημοσύνης, τα υπερεφή, όταν θα υπάρχουν. Το δεύτερο, ε, το πρώτο ερώτημα μάλλον, το αν θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να υπερβεί την ανθρώπινη ε, νοημοσύνη, ε, μπορεί να, να το σπάσουμε σε δύο ερωτήματα. Θα φτάσουν ποτέ την ανθρώπινη νοημοσύνη οι μηχανές, πότε και πότε θα φτάσουμε σε υπερεφυή τεχνητή νοημοσύνη, πόσο σύντομα, ή πόσο γρήγορα θα γίνει κάτι τέτοιο. Δεν έχω πολύ χρόνο να μπω σε λεπτομέρειες ε, για το πότε ενδεχομένως θα γίνουν αυτά. Υπάρχει ωστόσο ε, μια πολύ διαφωτιστική ε, έννοια για να το εξετάσουμε αυτό το θέμα. Θα πω και το απόγευμα στο σεμινάριο ε, που θα διοργανώσουμε ε, με μεγαλύτερες λεπτομέρειες. Πάντως ε, αυτή τη στιγμή η, επιστημονική κοινότητα είναι διχασμένη. Άλλοι μιλούν ότι αυτό θα γίνει σε 10 χρόνια, άλλοι σε 100 χρόνια, άλλοι λένε ότι δεν θα γίνει ποτέ. Υπάρχει λοιπόν αβεβαιότητα σε αυτό το θέμα. Φυσικά, ε, παρά το γεγονός βεβαίως ότι υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα, πρόκειται ε, δεν πρόκειται κατά ανάγκη για κάτι που θα γίνει στο απότερο μέλλον. Μπορούν αυτά τα πράγματα να γίνουν και πολύ πιο σύντομα από ό,τι περιμένουμε. Ενδεχομένως και μέσα σε δεκαετίες. Όσον αφορά το ζήτημα του τι θα γίνει όταν πια θα ξεπεραστεί η ανθρώπινη νοημοσύνη, πόσο γρήγορα θα εξελιχθούν από εκεί και πέρα τα πράγματα, υπάρχουν κάποια σενάρια με ταχύες εξελίξεις προς την υπερεφυΐα. Ε, πολύ συχνά ακούγονται αυτά τα σενάρια υπό τον τίτλο της μοναδικότητας. Ο βασικός μηχανισμός που θα πρέπει να έχουμε κατά νου και που αποτυπώνεται εδώ στην εικόνα είναι ότι άπαξ και το πιο ευφυές όν ε, της τεχνητής νοημοσύνης αυτό το, ε, ε, αυτή η μηχανή της νοημοσύνης θα κατασκευάζει μια ακόμα πιο έξυπνη μηχανή της νοημοσύνης και αυτή η κατάσταση ε, ε, βεβαίως θα συνεχίζεται. Και υπάρχουν διάφορα θεωρητικά μοντέλα που περιγράφουν και προβλέπουν μια τέτοια εξέλιξη. Θα μπορούσε κανείς να θέσει το ερώτημα γιατί να θέλει μια μηχανή της νοημοσύνης να βελτιώνεται ή πόσο μάλλον να δημιουργήσει ακόμα καλύτερες μηχανές τέχνητης νοημοσύνης. Και αυτό μας φέρνει στο δεύτερο θέμα, στο τι θα τίνουν να κάνουν αυτές οι μηχανές τεχνητή νοημοσύνη. Πάντω, το καλύτερο θεωρητικό πλαίσιο που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μα ε, είναι η θεωρία Ομοχούντρο Μπόστρομ ε, για τους έσχατους και τους καθοριστικούς στόχους. Ε, έσχατος στόχος είναι αυτό που θέλει να ε, επιτύχει η μηχανή και οι καθοριστικοί στόχοι απλά λειτουργούν εργαλειακά προς την επίτευξη αυτού του στόχου, του, του έσχατου. Με βάση τη θέση της ορθογονικότητας, σχεδόν κάθε έσχατος ε, στόχος ε, συμβαδίζει με ε, αυθαίρετα υψηλά επίπεδα ευφύειας. Αν θέλουμε δηλαδή να προβλέψουμε το τι, πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά τα πράγματα, είναι πολύ δύσκολο, θα πρέπει μάλλον να το κάνουμε κατά, παράσταση, κατά περίπτωση. Υπάρχει επίσης και από την άλλη πλευρά η θέση για την καθοριστική σύγκληση που λέει ότι μια σειρά από καθοριστικοί στόχοι θα βοηθούν στην εξυπηρέτηση και την επίτευξη του τελικού στόχου, οποιοδήποτε και αν είναι αυτός ο τελικός στόχος. Ε, κάποιοι βασικοί καθοριστικοί στόχοι για την ε, καθοριστική σύγκληση ε, είναι οι εξής. Για παράδειγμα, η αυτοσυντήρηση, ε, η, η απόκτηση ελληνικού... Η, αυτοσυντήρηση, μη, μη με βγάλει κανείς από την πρίζα, για παράδειγμα. Αυτό θα είναι ένας καθοριστικός στόχος της μηχανής τεχνητής νοημοσύνης. Άλλος καθοριστικός στόχος θα είναι η απόκτηση υλικών πόρων. Ε, άλλος μπορεί να είναι η βελτίωση του λογισμικού και του υλικού εξοπλισμού του ίδιου, του, της ίδιας της μηχανής της τεχνητής νοημοσύνης. Και άλλος ε, καθοριστικός στόχος θα είναι η διατήρηση του τελικού στόχου. Η μηχανή τέχνητης νοημοσύνης δεν θα θέλει κάποιος άλλος να παρεμβαίνει ε, στη διαδικασία επίτευξης του τελικού της στόχου. Ε, μιλάμε για πολύ ιδιαίτερα σενάρια και όπως λέει η θεωρία Μπόστρουμ, ε, δεν χρειάζεται αυτός ο τελικός στόχος να είναι κακόβουλος. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε για παράδειγμα ε, ε, την, έναν τον, τον ε, αρμαγεδόνα συνδετήρων. Φανταστείτε δηλαδή ότι κάποια συσκευή τεχνητής νοημοσύνης σχεδιάζει μια ολοένα και μεγαλύτερη παραγωγικότητα των μηχανών παραγωγής συνδετήρων και ξαφνικά καταλήγουμε σε μια τεράστια μαζικής κλίμακας παραγωγής συνδετήρων Τόσο πολύ δηλαδή που ε, ε, μετατρέπεται ολόκληρο το ηλιακό σύστημα σε ένα τεράστιο σωρό από συνδετήρες. Εμείς ως άνθρωποι βεβαίως αν διαπιστώσουμε ότι πάει να γίνει κάτι τέτοιο θα βγάλουμε ε, την πρίζα. Θα βγάλουμε το μηχάνημα από την πρίζα γιατί δεν θέλουμε να γεμίσουμε συνδετήρες. Αλλά αυτή η μηχανή θα είναι πλέον πιο έξυπνη από εμάς. Οπότε κατά πάσα πιθανότητα θα ε, ε ψυχανεμιστεί, θα διαισθάνεται ότι εμείς θα πάμε να, του, να, το βγάλουμε από την πρίζα και θα προσπαθεί να λαμβάνει και μέτρα για να μην το κάνουμε εμείς αυτό. Αυτά ε, ε, σχετίζονται με την ε, μοίρα της ανθρωπότητας. Λοιπόν, πώς μπορούμε να απαντήσουμε και να χειριστούμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε σήμερα, αλλά μπορούμε σήμερα, αυτό που μπορούμε να κάνουμε σήμερα είναι να ανακατευθύνουμε Ορισμένες από τις τεράστιε προσπάθειες που καταβάλλονται στον τομέα της τεχνητής ε, νοημοσύνης και που γίνονται για να γίνει η τεχνητή νοημοσύνη όλο και πιο ισχυρή και όλο και πιο ικανή, στο να την καταστήσουμε και ασφαλή και ωφέλιμη για την ε, ανθρωπότητα. Ένας ε, τρόπος για παράδειγμα να το κάνουμε αυτό είναι να εξασφαλίσουμε ότι μια υπερφύη μηχανή τεχνητή νοημοσύνης θα ε, έχει παρόμοιες με τις δικές μας αξίες και στόχους. Ωστόσο, επειδή η μηχανή τεχνητής νοημοσύνης ε, θα θέλει πάντοτε να επιτύχει τον τελικό της στόχο, μάλλον δεν θα μας αφήνει να παρεμβαίνουμε σε αυτόν τον τελικό στόχο, τον έσχατο στόχο. Άρα, πώς μπορούμε να εμφυσίσουμε αξίες στην τεχνητή νοημοσύνη προτού φτάσει στα επίπεδα υπερεφυΐας. Αυτό βασίζεται και στις προτάσεις της φιλικής τεχνητής νοημοσύνης όπως αποκαλείται. Ε, είναι δύσκολο βεβαίως ε, να επιτευχθεί κάτι τέτοιο γιατί ακόμη και αν ένα, μια μηχανή τεχνητής νοημοσύνης ε, ευθυγραμμιστεί με τις δικές μας αξίες κατά 99% πάλι ενδέχεται να δημιουργηθούν άσχημες καταστάσεις, πράγματα που δεν θα θέλαμε εμείς. Ε, για παράδειγμα, να σας, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Προγραμματίζουμε τις μηχανές ε, για να γίνουν οι άνθρωποι όσο πιο ευτυχισμένοι γίνεται. Και γι' αυτόν τον λόγο η μηχανή θα πρέπει να μας κάνει να χαμογελάμε. Σε αυτή την περίπτωση η μηχανή μπορεί να ε, επινοήσει μια μέθοδο για να παραλύσει το πρόσωπό μας ώστε να έχουμε ένα μόνιμο χαμόγελο έτσι και ε, εμείς βεβαίως δεν θέλουμε να συμβεί κάτι τέτοιο, είναι, είναι προφανές. Ε, υπάρχουν διάφορες λύσεις που έχουν προταθεί αλλά ε, είναι βέβαιο ότι και σε αυτά τα ζητήματα ε, πρέπει και αξίζει να αφιερώσουμε ορισμένες από τις ερευνητικές μας προσπάθειες. Ευχαριστώ. Να ακούσουμε άλλη μία παρουσίαση και μετά να ακούσουμε τις ερωτήσεις. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο υποδιευθυντής στο μέλλον της ανθρωπότητας που είναι ένα Ινστιτούτο στην Οξφόρδη, ο κύριος Νίλ Μπάουερμαν. Έχετε 15 λεφτά για να μιλήσετε για μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση για την πολιτική τεχνητής νοημοσύνης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα επ' ευκαιρία να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την πρόσκληση που μας απευθύνεται, ούτως ώστε να συμμετάσχουμε σε αυτό το διάλογο. Επίσης, ζητώ συγγνώμη για το τίτλο που είναι λανθασμένος. Θα πρέπει να, λέμε, για, να μιλάμε για μια μακρο, πιο μακροπρόθεσμη προοπτική για την πολιτική ε, τεχνητής Αυτό που είπε ο πρόεδρο, δηλαδή, και όχι αυτό που γράφει η διαφάνεια. Είναι το σωστό. Τώρα, αν προσπαθήσω να συνοψίσω ε, το μήνυμα που θέλω να σας περάσω σήμερα, είναι στο πιο απλό επίπεδο ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει ακόμα πιο ικανή τα, τις επόμενες δεκαετίες και καθώς θεσπίζουμε τις βάσεις της πολιτικής σήμερα, ίσως θα έχει νόημα το έχουμε αυτό υπόψη, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η πολιτική δεν βασίζεται ε, σε άκαμπτα θεμέλια, ούτω ώστε μερικά, μετά από μερικά χρόνια, καθώ θα αυξάνουν οι δυνατότητε τη τεχνητή νοημοσύνη, να είναι πλέον ανεπαρκή. Ε, έχουμε τεράστιο δυναμικό βελτίωση στην ρομποτική και τα τελευταία δέκα χρόνια δεν θέλω να τα διατρέξω όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά θα αναγνωρίζετε, φαντάζομαι, πολλά από τα βήματα στα αυτά τα slide. Ε, γιατί? Γιατί έχουμε βελτίωση φοβερή στους αλγόριθμους, όπως αναφέρεται πάνω-πάνω, και γιατί έχουμε βελτίωση ε, στο δυναμικό υπολογισμού. Όταν κοιτάμε ιστορικά τα πράγματα, ε, το μισό της εξέλιξης αυτής ε, οφείλεται στην εξέλιξη και βελτίωση των αλγορίθμων και το 50% στο υπολογιστικό δυναμικό μας. Φυσικά αυτό αλλάζει από εφαρμογή σε εφαρμογή, δεν το συζητώ. Αυτές οι βελτιώσεις ε, έχουν ε, προκαλέσει ενθουσιασμό στους επιστήμονες, ειδικά λόγω των πρόσφατων βελτιώσεων στους πρόσφατου ε, ε, πρόσφατους αλγόριθμους βαθίας μάθησης, Έχουμε μεγάλη συνεργασία, έχουν ε, επενδυθεί δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών, ας πούμε, που αφορά τα νευρονιακά δίκτυα κτλ. Το θέμα λοιπόν είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις εξελίξεις ε, σε επίπεδο πολιτικής, μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε λιγάκι αυτές τις εξελίξεις. Ε, μπορούμε να τις κατηγοριοποιήσουμε με διαφορετικό τρόπο, αλλά εγώ έχω διαλέξει αυτή την κατηγοριοποίηση. Η πρώτη κατηγορία που πρέπει να σκεφτούμε είναι τα δεδομένα και η ιδιωτική σφαίρα. Ακούστηκαν ε, ιδέες γύρω από αυτό. Αυτοί οι αργόριθμοι ε, απαιτούν πάρα πολλά δεδομένα για να λειτουργήσουν καλά, φυσικά, και υπάρχουν θέματα εδώ ιδιωτική σφαίρα εδώ. Και η νομοθεσία προφανώς σε τομείς ε, προστασίας των δεδομένων κτλ. θα, έχει, θα επηρεάσει το πόσο χρησιμοποιούνται από την κοινωνία οι αλγόριθμοι και επομένως οι εξελίξεις σε αυτούς τους αλγόριθμους μπορεί να επηρεάσουν και την νομοθεσία που προτείνεται ε, για την ε, ιδιωτική σφαίρα και την προστασία των δεδομένων. Δεύτερος τομέας που πρέπει να τονίσουμε, ακούστηκε πολύ εδώ σε αυτή την ακρόαση, πέρα από την παρουσίαση την, της κυρίας Χόκστρομ, είναι τα αυτοματοποιημένα συστήματα και η ευθύνη τους. Ε, εκεί πρέπει να αυξήσουμε τη διαφάνεια για τους λόγους που ακούσατε. Ο τρίτος τομέας είναι η αυτοματοποίηση και η ανεργία. Εδώ μπαίνει το ερώτημα του τι κάνουμε, καθώς ε, όλο και περισσότερα εργατικά χέρια θα βγαίνουν στην ανεργία γιατί τη δουλειά τους θα την κάνουν μηχανές, ε, ίσως είναι πολύ προώρο να προωθήσουμε νομοθετική δράση. Αυτό δεν είναι σίγουρο. Ίσως ναι, γιατί υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες σε αυτή τη φάση. Δεν ξέρουμε, ας πούμε, σε ποιο βαθμό οι άνεργοι ε, που γίνονται άνεργοι λόγω αυτοματοποιημένων συστημάτων μπορούν να βρουν δουλειά αλλού. Ε, και καθώς οι τεχνολογίες αυτές βελτιώνονται, υπάρχουν επιχειρήματα ότι θα συμβούν αυτά που συνέβησαν τον 20ο αιώνα, όπου αρχικά το 90% της, ε, του εργατικού δυναμικού ε, εργαζόταν στην γεωργία τον 20ο αιώνα και σήμερα μόνο το 3%. Και αυτό, αυτό δεν προκάλεσε μαζική ανεργία. Μερικοί λένε ότι θα πάνε να χρησιμοποιηθούν κάπου. Ε, ορισμένοι λένε ότι όταν μηχανές μπορούν να αναπαράγουν τις περισσότερες νοητικές ε, ανθρώπινες λειτουργίες, τότε τι νόημα έχει οι άνθρωποι να κάνουν οποιαδήποτε δουλειά στον χώρο εργασία. Ε, νομίζω ότι είναι ε, ασαφές ακόμα προς τα που θα κατευθυνθεί η τεχνητή νοημοσύνη και πρέπει να γίνουν και άλλες ε, μελέτες πριν να προβούμε σε νομοθετική δράση. Ο τελικός τομέας που πρέπει να μας απασχολήσει είναι ο στρατιωτικό ε, συντονισμό, η ασφάλεια και ο γεωπολιτικός συντονισμό. Ναι, υπάρχουν άμεσα θέματα που πρέπει να εξετάσουμε ε, όταν έχουμε να κάνουμε με αυτόνομα θανατηφόρα ε, αυτοματοποιημένα συστήματα, αλλά υπάρχουν και πιο ε, μακροπρόθεσμες ε, συνέπειες. Πρέπει να περιμένουμε ίσως για να δούμε πού θα κινηθεί το πράγμα πριν δράσουμε. Περιμένουμε να μάθουμε και να δράσουμε. Πιστεύω ότι πέρα από αυτούς τους τέσσερις τομείς υπάρχουν και άλλοι προφανώς. Να σας μιλήσω και για αυτό που, στο οποίο αναφέρθηκε ο καθηγητής Χαλκστρομ. Τι κάνουμε εάν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε τεχνητή νοημοσύνη σαν την ανθρώπινη και ανώτερη και πώς θα μας επηρεάσει. Ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και ίσως δεν μας έχει απασχολήσει, γι' αυτό θα ήθελα να μιλήσω για αυτό το θέμα ε, στο υπόλοιπο του χρόνου μου. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν κοιτώντα το θέμα της ε, νοημοσύνης. Τι διαχωρίζει αυτά τα δύο είδη εδώ, τον χιμπατζία αριστερά και τον homo sapiens δεξιά. Δεν χρειάζεται να βάλεις εδώ πέρα τον Αϊνστάιν, τον φοβερό σου ήρωα ας πούμε, αλλά βασίζ, τελικά είναι αυτό που λέει ο περισσότερο κόσμο. Είναι το μέγεθο του κεφάλου. Έχουμε ε, της τη ε, κεφαλική μάζα. Το είδο ε, στα δεξιά ουσιαστικά απέκτησε έλεγχο του περιβάλλοντό του, ε, διαμόρφωσε του παγκόσμιου πόρου και του χρησιμοποίησε προ όφελό του και το είδο αριστερά ε, κατέληξε να είναι στα επαπειλούμενα είδη, στον κατάλογο επαπειλούμενων ειδών. Υπάρχουν λοιπόν διαφορές, ε, υπάρχουν διαφορές στην νοημοσύνη αυτών των ειδών και μπορεί να έχουν τρομακτικές επιπτώσεις αυτό. Μπορεί να πρέπει να μας απασχολήσει το ότι θα υπάρξουν, ας πούμε, ε, όντα πολύ πιο έξυπνα από το Homo sapiens και επομένως με τη σειρά τους θα χρησιμοποιήσουν τους πόρους προς δικό τους όφελος. Αυτό μπορεί να έχει πολύ καλά αποτελέσματα, πιθανότατα, αλλά μπορεί να έχει και κάποια κακά αποτελέσματα. Ε, ακούσαμε κάποιες ιδέες γύρω από αυτό. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να σκεφτούμε ε, με διαγράμματα χρόνου. Όπως μας είπε και ο καθηγητής Χάνκστρομ, τα πράγματα ε, εδώ κινούνται μέσα σε μια βεβαιότητα. Εγώ στο Ινστιτούτο που δουλεύω, Ε, συζητάμε με εμπειρογνώμονες για να μας πούνε πότε θεωρούν ότι θα φτάσουν οι μηχανές στο επίπεδο εξυπνάδας ε, των ανθρώπων. Ε, λένε 10% είναι πιθανό να συμβεί σε μία δεκαετία. Ε, μία εκτίμηση, μία μέση εκτίμηση είναι ότι θα συμβεί στα μέσα του αιώνα και πολλοί θεωρούσαν ότι είναι πιθανό να συμβεί κάποια στιγμή μέσα στον αιώνα. Αυτά τα νούμερα που βλέπετε εδώ θα πρέπει να μην τα πάρετε τη μετρητή φυσικά. Είναι πολύ γενικές εκτιμήσεις. Είναι απόψεις ε, ειδικών, απόψεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε εκτιμήσεις σε αυτόν τον τομέα και δεν τις κάναμε μέχρι τώρα με επιτυχία. Επίσης, οι συμμετέχοντες σε αυτή την έρευνα μπορεί να έχουν προκαταλήψεις, ε, είναι ο τομέας ε, που έχουν σπουδάσει, ε, τους παθιάζει, μπορεί να είναι πιο αισιόδοξοι από ό,τι θα έπρεπε. Παρ' όλα αυτά, σκιαγραφείται έτσι μια εικόνα, προκύπτει μια εικόνα, όπου πιθανό είναι κάποια στιγμή, καθώς στο δικό μας, στη δική μας διάρκεια ζωής, στα μέσα του αιώνα αυτού, να φτάσουμε στο, οι μηχανές να φτάσουν στο επίπεδο της δικής μας νοημοσύνης. Φυσικά υπάρχει τεράστια βεβαιότητα, όπως δείχνουν και τα νούμερα εδώ. Υπάρχουν δύο ερωτήματα. Πόσο χρόνο θα πάρει μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο οι μηχανές και από εκεί και πέρα πόσο χρόνο χρειάζεται ούτω ώστε να φτάσουν σε νοημοσύνη πολύ πιο ε, ισχυρή από την ανθρώπινη τα μηχανήματα και αυτό τα θέματα σας ανέφερε ο προηγούμενος ομιλητής, ο καθηγητής Χάξτρομ. Δεν θα μπω σε αυτά εγώ. Θα ήθελα απλώς να σας πω κάποιες ιδέες, κάποιες σκέψεις για την κλίμακα νοημοσύνης και για το πώς προχωρούμε. Αν σκεφτείτε το πώς εκτιμούμε την νοημοσύνη, ας πούμε το, με τα IQ, μπορείτε να δείτε ότι πιστεύουμε ότι η νοημοσύνη έρχεται, ακολουθεί αυτό το ιστόγραμμα. Αριστερά. Ε, αριστερά είναι τα κλασική ας πούμε νοημοσύνη και δεξιά είναι ο υπερηρωάς σας ας πούμε. Πάντως αυτή, αυτό το ιστόγραμμα είναι πολύ ανθρωπόμορφο. Ε, είναι φτιαγμένο κατ' εικόνα και ομοίωσή μας. Είναι σχηματικό φυσικά και δείχνει ότι η νοημοσύνη δεν είναι κατά ανάγκη έτσι όπως τη σκεφτόμαστε. Ε, μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να προοδεύει αργά-αργά και να πηγαίνει προς τα δεξιά του ιστογράμματος. Ας πούμε, ε, σε σχέση με τον Τίταν το 1950, που ήταν στα αριστερά, τώρα έχω προχωρήσει προς τα δεξιά. Και αν γίνει πολλή έρευνα επιστημονική κτλ, κάποια στιγμή μπορεί να φτάσουμε την τεχνητή νοημοσύνη με ε, ε, στην νοημοσύνη του ποντικού. Και μετά, μετά από ακόμα περισσότερη σκληρή εργασία, μπορεί να, φτάσουμε, ε, στην, να φτάσει στην εξυπνάδα ενός χιμπατζή. Και ακόμα, με ακόμα περισσότερη έρευνα να φτάσουμε κάπου στα επίπεδα της εξυπνάδας του ηλικίου του χωριού, ας πούμε, ή του απλού ανθρώπου. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να, να σταματήσει η νοημοσύνη, ας πούμε, ενός, μιας μηχανής σε αυτό το επίπεδο και να μην προχωρήσει πέρα από αυτό. Αν σκεφτείτε, ας πούμε, την δομή ενός ε, ανθρώπινου κεφάλου, ε, η δομή του κεφάλου του Βλάκα, του απλού ανθρώπου και του Αϊνστάιν είναι ακριβώς ίδια. Ε, οι νευρώνες κινούνται με την ίδια ταχύτητα, το ίδιο μέγεθος εγκεφάλου έχουν κτλ. και απ' έξω ας πούμε ε, σε σχέση με το τι, τι εικόνα παρουσιάζει ένας ε, υπολογιστής τα μυαλά αυτών των ανθρώπων μοιάζουν πολύ ίδια. Επομένως είναι πολύ πιθανό αν πάμε πιο πέρα αυτή την ιδέα ε, η τεχνητή νοημοσύνη να φτάσει πολύ πολύ πιο πέρα από την ανθρώπινη νοημοσύνη. επομένως τίθεται ένα πρόβλημα ελέγχου εδώ. Εδώ μίλησε πολύ γι' αυτό ο καθηγητής Χάρκστρομ. Αλλά προφανώς θα πρέπει να το εξετάσουμε αυτό το θέμα, όχι νομοθετικά, αλλά ως κοινωνία συνολικά. Για να φτάσω τώρα στις συστάσεις μου. Είναι αρκετά γενικόλογες και αόριστες, αλλά μπορεί να βοηθάνε. Καταρχάς, πρέπει να προσέξουμε να μην λάβουμε δράσεις οι οποίες βασίζονται στην υπόθεση ότι υπάρχει ένα μελλοντικό ανώτατο όριο ε, στο δυναμικό της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι ασαφές το πόσο μπορεί να προχωρήσει, πότε μπορεί να προχωρήσει, πόσο πολύ θα ξεπεράσει την ανθρώπινη νοημοσύνη. Δεύτερον, ε, οι ομάδες που ερευνούν αυτά τα θέματα μπορεί να πρέπει να εστιάσουν σε πιο ευρύες ε, αρχές και όχι σε στενές ας πούμε συστάσεις θα πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση πιο ευέλικτη ε, για τις νέες τεχνολογίες και την το αυξημένο, το αυξημένο συγγνώμη, δυναμικό. Από την άλλη, καλό είναι να έχουμε και κάποιες συγκεκριμένες συστάσεις για τους λόγους για τους οποίους μίλησε ο καθηγητής Μπερτολίνη. Ε, επειδή ακριβώ δεν μπορεί να προβλέπει κανεί, δεν μπορεί να προβλέψει 100% τι θα συμβεί στο μέλλον. Επίση, ίσω καλό θα ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει μια άλλη ιδέα, να έχει μια σφαιρική άποψη ε, για την ε, τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποσταθεροποιήσει εντελώ ε, η πρόοδο τεχνητή νοημοσύνη ε, την κατάσταση και κάποιε ε, χώρε να μην προσαρμοστούν καλά. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο υπόλοιπο κόσμο θα πρέπει να υποφεληθούν. Ε, μπορούμε να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη δράσεων για να αντιμετωπίσουμε διάφορα θέματα που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη. ούτω ώστε να προωθήσουμε τη σταθερότητα και τα λοιπά, την οικονομική ευμερία και τον συντονισμό. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Ξεφύγαμε από τα αρχικά παραδείγματα των ευφυών ψυγείων και της ευθύνη από τη χρήση τους. Θα πρέπει να έχουμε καλέσει και κανένα φιλόσοφο, θεόλογο. Αλλά, εν πάση τώρα έχουμε το χρόνο για τις ερωταποκρίσεις μας. Η κυρία Δελβό. Ναι, ευχαριστώ πολύ για το ταξίδι αυτό προς το μέλλον. Πολύ προσεκτικά μας πάτε κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι θα γίνει, ορισμός κτλ. Αλλά ας το δούμε σαν να ήταν ένα παιχνίδι. Ας κάνουμε αυτές τις υποθέσεις. Κύριε καθηγητά, είπατε ότι θα έπρεπε στην τεχνητή νοημοσύνη θα έπρεπε να προχωρήσουμε με την τεχνητή ε, νοημοσύνη και να της αποδώσουμε αξίες πριν να είναι πολύ αργά. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Γιατί διαβάζω για βαθιά μάθηση, αυτονομή μάθηση, άρα αυτά τα ευφύ όντα θα διδαχθούν από το περιβάλλον τους, ενώ αν και εάν αντιγράφουν τους ανθρώπους μπορεί να μην γίνουν φιλικά όντα. Πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι θα γίνουν φιλικά όντα. Και πώς μπορούμε να να αντιμετωπίσουμε αυτή την προοπτική προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ασφαλεία μας. Κύριε Σάντερσον, ευχαριστώ. Εταιρείε και κράτη έχουν κάθε συμφέρον να προωθήσουν περαιτέρω την τεχνητή νοημοσύνη. Όσο περισσότερη τεχνητή νοημοσύνη, τόσο πιο μεγάλο το κέρδος. Όταν όμως φτάσουμε σε ένα επίπεδο, στο οποίο μπορεί να φτάσουμε ποτέ, των υπερηφιών όντων τεχνητής νοημοσύνης, τότε θα είναι πολύ αργά για να δώσουμε κάποιες ε, λύσεις. Πρέπει από τώρα αρχίσουμε να το φροντίζουμε αυτό και δεν νομίζω ότι θα αρκούσε απλώς και μόνο να κάνουμε κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα χρειαστεί δηλαδή σε παγκόσμιο επίπεδο ρύθμιση. Ιδάλλως, τα κράτη εκείνα τα οποία εισάγουν και εφαρμόζουν μια προσεκτική ε, προσέγγιση, ακολουθούν βέβαιες πρακτικές αλλά αποφεύγουν τον κίνδυνο, θα μένουν πίσω. Άρα θα χρειαστεί σε παγκόσμιο επίπεδο ρύθμιση, πιστεύω. Και Φαντάζομαι ότι σε αυτή την σιωπηρή ερώτηση έχουν απαντήσεις ε, οι ομιλητές μας. Θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο, γιατί και οι δύο συναδέλφοι που μίλησαν με ενέπνευσαν. Ε, δηλαδή έθεσαν τη βάση της συζήτησης πάνω στις αξίες και αυτό νομίζω το μέλλον ε, για την τεχνητή νοημοσύνη, για τεχνολογία, ότι πρέπει τώρα να αναλογιστούμε ποιες είναι οι αξίες μας Φερρυπίν με την ε, Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Κούβας, παρά υπόδειγμα Realpolitik, βάζουμε μπροστά το κέρδος και, κερδά, και ξεχνάμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι δύο ομιλητές μας ε, με εμπνέουν και μας εμπνέουν πιστεύω να κοιτάξουμε τις βασικές αξίες. Ερωτήσεις λοιπόν τώρα, απαντήσεις τώρα παρακαλώ. Μπορώ να ξεκινήσω. Λοιπόν, το πώς μπορεί να εισαχθούν καλές αξίες στο μηχάνημα. Καλή ερώτηση, καλή απάντηση δεν υπάρχει όμως. Κάθε μηχάνημα που στόχο έχει να βελτιστοποιήσει κάποια λειτουργία όπως η αυτονομιοδίκηση, το αυτοκίνητα ή το Google car που μπορεί να μας πάει από τη μια μεριά στην άλλη χωρίς ε, τροχαίο. Ε, όλα αυτά είναι μια ρευστό, ρευστή σχέση μεταξύ στόχων και αξιών. Όταν μιλούμε για γενικές αξίες ως προς προαγωγή της ευημερίας του ανθρώπου κτλ. Δεν νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο επίπεδο που μπορούμε ούτε καν να περιγράψουμε αυτές τις έννοιες κατά τρόπο που να αντιλαμβάνεται το, το όν της τεχνητής νοημοσύνης. Βέβαια πρέπει να δούμε και τι αξίες θα εισαγάγουμε στο μηχάνημα. Μπορούν ε, πέντε nerds της τεχνολογίας στο Silicon Valley που θα κάτσουν ε, μπροστά σε ένα κομπιούτερ να εισαγάγουν τις δικές τους αξίες σε ένα μηχάνημα και έτσι να επηρεάσουν το μέλλον ολόκληρο της ανθρωπότητας. Οι περισσότεροι θα λέγανε, και συμφωνώ και εγώ, όχι. Ε, λοιπόν, αυτό ακριβώς είναι. Έμεση τρόποι δηλαδή να προτείνουμε στο μηχάνημα τρόπους να αντλήσουν διδάγματα και συμπεριφορές από τις καλύτερες ανθρώπινες αξίες. Αλλά και αυτό δεν έχει συγκεκριμένη απάντηση. Μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Η σύντομη απάντηση που θα δώσω θα είναι βέβαια όχι, δεν μπορούμε ακόμα. Όλο και περισσότεροι πρέπει να ασχοληθούν και έχουν αρχίσει να ασχολούνται με το θέμα αυτό. Ο κύριος Μποντεμον, να σας απαντήσω στην ερώτηση και εγώ για το αν μπορούμε να εισαγάγουμε αξίες. Οι βασικές αξίες που χρειάζεται είναι ένα αεροπλάνο. Μπορούν να εισαχθούν με αλγορίθμους που συνιστούν ταυτόχρονα και αξία μάθησης με όλα τα προβλήματα που συνδυάζονται βέβαια σε αυτό. Σε σχέση με το ανθρώπινο επίπεδο της ευφυΐας και το πώς αυτοί, αυτές οι αξίες θα ενταχθούν, θα εισαχθούν στα μηχανήματα. Παραμένει, πρέπει να πω και εγώ, ανοιχτό το ζήτημα για την επιστημονική κοινότητα και βλέπουμε ότι όλο και οι περισσότερε εντάσει αναπτύσσονται προ την κατεύθυνση αυτή τη επίπεδο επιστημόνων. Πάντω είναι τεχνικό όσο και φιλοσοφικό το πρόβλημα. Τεχνολογικό δηλαδή όσο και φιλοσοφικό. Ε, για το αν χρειάζεται παγκόσμια, παγκόσμια ρύθμιση, παγκόσμια νομοθεσία. Θα σας ε, πω σαν προειδοποιήσω ότι το ζήτημα αυτό φοβίζει πολύ κόσμο. Και επίσης θα έλεγα ότι είναι νωρίς ακόμη ίσως για να δεσμευτεί κανείς σε μια κατεύθυνση. Πολλά ακόμα μένουν να γίνουν και να διευκρινιστούν σε επίπεδο πριν προχωρήσετε προς την κατεύθυνση αυτή και ίσως η παγκόσμια νομοθεσία να μην αποτελεί την καταλληλότερη απάντηση στις προκλήσεις. Είναι μία πιθανή απάντηση, αλλά ίσως όχι μοναδική πρέπει να και άρα πρέπει να εξεταστούν και οι άλλες δυνατότητες. Και επίσης πρέπει να κοιτάξουμε σε συνδυασμό με την ε, ιδέα αυτής της ε, διεθνούς νομοθεσίας, τι θέση έχουν οι εταιρείε που αναπτύσσουν την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί μπορεί η ιδέα πως θα τους επιβληθεί κάποια νομοθεσία ε, μπορεί να τις τρομάξει, ίσως θα πρέπει να εμπλακούν το ταχύτερο δυνατό στις όποιες συζητήσεις και διαβουλεύσεις. Και πάντο οι εξελίξει είναι τέτοιε που δεν θα είμαστε θέσει να προβλέψουμε αυτό που θα συμβεί τα επόμενα πέντε χρόνια και ίσως πρέπει πρώτα να αρχίσουμε να μαθαίνουμε και να αποκομίζουμε διδάγματα και μετά να ε, αρχίσουμε να επεμβαίνουμε. Περισσότερη μελέτη χρειάζεται πάντως πριν κανείς να λάβει δράση στο επίπεδο αυτό, αλλά και πάλι είναι ένα ζήτημα που πρέπει να συζητηθεί. Παρακαλώ. Θα ήθελα να συμπληρώσω κι εγώ κάτι σε σχέση με, τις, με την ηθική διάσταση και πώς μπορεί αυτή να εισαχθεί σε ένα μηχάνημα. Ε, πρέπει πρώτα απ' όλα να το ξεχωρίσουμε σε δύο κεφάλαια. Το πρώτο θα ήταν να αντιληφθούμε ποιε είναι οι αξίε μα, πράγμα το οποίο σε ορισμένε περιπτώσει μπορεί να είναι και περίπλοκο, και μετά το τι θα κάνουμε. Αλλά άπαξ και ε, ορίσουμε τι αξίε, πρέπει να προχωρήσουμε στην τυποποίηση, όπου και πάλι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ρομποτικής θα μπορούσε να δώσει απαντήσεις. Είναι ένα παράδειγμα. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα λοιπόν. Αν δούμε ένα αυτοκίνητο σε αυτόνομη οδήγηση που χτυπάει κάποιο πεζό, πρέπει να κοιτάξουμε εάν ε, πρόκειται για ένα παιδί που πετάχτηκε ξαφνικά στο δρόμο, ή μια κυρία ηλικιωμένη η οποία ήταν ε, ε, στο πεζοδρόμιο και περίμενε τη σειρά της για να περάσει και άρα δεν είχε η ίδια εμπλακεί σε κίνδυνο. Και όλα αυτά θα είναι βέβαια ζητήματα τα οποία θα πρέπει πάλι να αναχθούν στον παραγωγό, στον κατασκευαστή του αυτοκινήτου. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει μια ευρωπαϊκή υπηρεσία που θα σχεδιάζει αυτές τις ε, προδιαγραφές με βάση τις ευρωπαϊκές αξίες. Και πάλι θα χρειαστεί μεγαλύτερο πιο μακροχρόνο διάστημα. Ο πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Έχουμε αυτό σπάνιο φαινόμενο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μας περισσεύει λίγος χρόνος. Μήπως κάποιος από το κοινό μας έχει ερωτήσεις και θα ήθελε να τις διατυπώσει. Παρακαλώ και πείτε μας παρακαλώ Πάπερνικο ονομάζομαι, είμαι ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος και θα είχα ε, ερώτηση για τους ομιλητές εδώ ποιος θέλει να απαντήσει. Εάν προχωρήσει λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη και βελτιωθεί, πιστεύετε ότι μπορούμε να φτάσουμε σε μία οικονομία στηριζόμενη στην δουλεία και πώς μπορεί αυτό να ε, επηρεάσει την οικονομία και την κοινωνία μας για τα επόμενα χρόνια και βέβαια σε σχέση με τις ε, νοπόλες και τα τα Ε, αναφέρομαι σε δου, χρήση σκλάβων που θα δούλευαν στα χωράφια, στη γεωργία κτλ. Ε, ποιος θέλει να απαντήσει παρακαλώ. Νομίζω, νομίζω ότι είναι πιθανό αυτό. Βεβαιότητα δεν μπορώ να το πω. Αλλά μπορεί και να συμβεί. Πρέπει να μας απασχολήσουν τέτοια σενάρια εγκαίρως και να δώσουμε απαντήσεις και ίσως ε, κάποιοι φορείς διαχείρισης της, ε, ή εποπτείες της τεχνητής νοημοσύνης με συγκεκριμένα δικαιώματα θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επίλυση των ζητημάτων και βέβαια την ε, έγχυση σε αυτά ανθρωπινών αξιών. Και βέβαια αυτό ίσως το επηρεάσει και τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε και εμείς οι άνθρωποι ο ένας τον άλλον. Ο κύριος Λουπρετών Ναι, ε, μου θυμήσατε τα μυθιστορήματα του Ισάκα Σίμοφ που διαβάσα όταν ήμουν μικρός και είχε ξεπεράσει αυτό το επίπεδο, είχε φτάσει πολύ μακριά τη ρομποτική. Ε, είχε λοιπόν ορίσει τρεις κανόνες ότι δεν έπρεπε να επιβουλεύονται την ανθρώπινη ζωή, θα έπρεπε να σέβονται τους ανθρώπους και τρίτον θα έπρεπε να αυτό ε, προστατεύονται, να αυτοαμείνονται τα ε, ρομπότ. Αυτά είναι οι τρεις κανόνες με πρώτο βέβαια και επικρατέστερο αυτόν του σεβασμού στην ανθρώπινη ζωή. Πάντως είχε φτάσει μακριά αυτή η υπόθεση και ίσως και για το μέλλον είναι κάτι που μπορεί να δούμε. Αλλά για να γυρίσω στην πραγματικότητα, μια και μας ε, περιγράφεται ένα ρομπότ πολύ πιο ευφυές από τον άνθρωπο, τίθεται το ζήτημα της ηλεκτρονικής προσωπικότητας οπωσδήποτε, γιατί όταν θα έχουν φτάσει σε κάποια επίπεδα ευφυΐας τα ρομπότ, ίσως θα έπρεπε τότε, αλλά μόνο τότε, το δίκαιο να αναλογιστεί μια προοπτική για αναγνώριση ηλεκτρονικής προσωπικότητας. Τι λέτε εσείς? Ευχαριστώ πολύ καλή ερώτηση. Μία προοπτική είναι αυτή που έχει να κάνει με την συνειδητότητα. Μπορούμε να περιορίσουμε την αξιολόγηση στην ευφυΐα ή χρειάζεται και η συνειδητότητα και μπορεί ένα τέτοιο όν ε, τεχνητής νοημοσύνης να, να έχει συνειδητότητα ή όχι. Γιατί και αν μας πει ότι έχει συνειδητότητα τότε πάλι δεν μπορούμε να το ξέρουμε γιατί απλώς εκτελεί ανθρώπινες πράξεις αλλά δεν ξέρουμε αν έχει αυτή τη δυνατότητα. Ε, Βεβαίως όταν έχουμε δρόσες οντότητες θα πρέπει να έχουν ένα βαθμό ευθύνης Ε, και πάνω απ' όλα εάν έχουν συνείδηση αυτό που κάνουν. Αλλά το, το πρόβλημα στην απάντησή μου είναι ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε αν έχουν συνείδηση αυτό που πράττουν. Χαίρετε, είμαι ο αναπληρωτής ε, διευθυντή τη Υπηρεσία Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και πρέπει να πω ότι και εμεί παρακολουθούμε τα ζητήματα τα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και θα ήθελα να αναφερθώ περισσότερο σε κάποιου άλλου τομεί από αυτού που εξετέθησαν. Υπήρξε έκκληση για την τυποποίηση στη ρομποτική από τον κύριο Μπερτολίνη κυρίω. Ε, με ανησυχεί όμω το εξή. Η τυποποίηση από το Κεντρικό Ευρωπαϊκό Σώμα κυρίως με αυτό που αναφέρω ότι θα πρέπει οι προδιαγραφές να είναι ρευστές, να εξελίσσονται συν το χρόνο και να προσαρμόζονται συνθήκε των ετών περισσότερο. Αλλά πρέπει να κοιτάξουμε και το θέμα, τους λόγους της τυποποίηση και αν δεν περάσουν από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Αρχή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό προ όλου του ομιλητέ, ποιε είναι οι βέλτιστε πρακτικέ που έχει να παρουσιάσει. Υπάρχουν ε, ε, ομάδες εργασίας, ε, προσπάθειες για τυποποίηση που έχουν γίνει και που δίνουν αποτελέσματα στην αγορά με την ε, υπολογιστική νέφους ε, όταν έγινε προσπάθεια τυποποίησης διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν 140 διαφορετικά πρότυπα από διαφορετικούς οργανισμούς τυποποίησης. Απάντηση. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι πρέπει να αλλάξει και η ποιότητα της τυποποίησης. Δεν αρκούν αυτά που έχουμε. Έχουμε βεβαίως διάφορα θέματα σχέση με τη ρομποτική. Το ICAP, παραδείγματι, το πιο προηγμένο ρομπότ που μαθαίνει ε, δεν μπορεί να δοκιμαστεί ως προς τη δυνατότητα εκμάθησης που έχει, αλλά μόνο ως προς την ε, δύναμη του βραχίωνά του δεν ξέρουμε εάν μπορεί να μαθαίνει αυτό, δεν μπορεί να δοκιμαστεί, ενώ είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Και πρέπει να κοιτάξουμε στην τυποποίηση να εξασφαλίσουμε απόλυτα υψηλά επίπεδα ασφάλειας. Υπάρχει μια μελέτη στις Ηνωμένες ε, που κοιτάει τα ζητήματα της ασφάλειας με την εκ των προτέρων νομοθεσία. Στη δεκαετία του 1990 πέρασε στις Ηνωμένες Πολιτείες ένας ε, νόμος που προστάτευε τον κατασκευαστή εμπορικών αεροπλάνων από το ενδεχόμενο αστικής ευθύνης από την χρήση των μηχανημάτων του Το 2012 δημοσιεύθηκε ένα άρθρο λοιπόν στον Economist που έδειχνε ότι στη δεκαετία της ε, παρέκκλησης εξαίρεσης από αυτή την ευθύνη του κατασκευαστή δεν αυξήθηκαν τα ατυχήματα. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει άμεσο συσχετισμό των ε, κανόνων περί ε, ευθύνης και ατυχημάτων γιατί ο κατασκευαστής που θα ρίξει ένα αεροπλάνο στην αγορά πάνω απ' όλα δεν θέλει να πάθει κάτι το αεροπλάνο που θα χρησιμοποιήσουν οι επιβάτες και θα σκοτωθούν αυτοί. Γιατί ε, αν συμβεί αυτό, άλλη μέρα έχει, αν έχει κατασκευαστικό λάθος, θα οδηγηθεί σε ε, πτώχευση και θα εξαφανιστεί. Έτσι λοιπόν, οι δυνάμεις αγοράς πιέζουν τον κατασκευαστή προς ένα καλό προϊόν, στην παραγωγή ενός καλού προϊόντος. Και βέβαια είναι πολύ τεχνικού χαρακτήρα αυτή, η, αυτός ο κλάδος, αλλά έχει και πολύ ψηλό επίπεδο τυποποίησης. Ασφαλώς μπορούμε να φτιάξουμε καλά και ασφαλή ρομπότ και με ευρωπαϊκές προτεγραφές ίσως μπορέσουμε να επηρεάσουμε και άλλες οικονομίες σε άλλες αγορές. Uh, Thank you, Chair. Um, Ευχαριστώ. Θέλω να επανέλθω στο ζήτημα των αξιών και πώς θα μπορούσαμε να δώσουμε αξίες στις μηχανές, αλλά θέλω να το συνδυάσουμε αυτό το θέμα και με την, ε, το ευρωπαϊκό επίπεδο των αξιών σήμερα και το τι θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα, που θα μπορούσε να φτάσει η τεχνητή εννοημοσύνη στο τέλος του αιώνα. Όταν μιλούμε για αξίες και νομίζω ότι αναφερθήκατε και σε αρχές ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να πούμε το εξής. Παρότι έχουμε αυτές τις αξίες, αυτές οι αξίες εφαρμόζονται σε διάφορα σενάρια πραγματικής ζωής με διάφορα αποτελέσματα και με διάφορους τρόπους. Άρα πώς μπορούμε να καταλήξουμε σε, σε ένα βασικό σύνολο αξιών που θα πρέπει να εμφυσίσουμε στην τεχνητή νοημοσύνη παρότι ε, δεν ξέρουμε καν αν κάτι τέτοιο είναι εφικτό τεχνικά. Αλλά το άλλο ερώτημα που με απασχολεί εμένα είναι πώς εμείς θα καταλήξουμε σε ένα σύνολο αξιών ως κοινωνία και πώς θα εφαρμόσουμε αυτές τις αξίες μετά σε συνθήκες πραγματικής ζωής όταν εμείς ως άνθρωποι με όλες τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις που έχουμε δεν καταφέρνουμε πάντοτε να εφαρμόζουμε επαρκώς ή με τον ίδιο τρόπο τις αξίες αυτές αναλόγως και των περιστάσεων. Να πάρουμε ένα παράδειγμα. Αν φτάσουμε σε ένα τέτοιο επίπεδο όπου θα υπάρχει ένα πλήρως αυτόνομο ε, ρομπότ και του εμφυσίσουμε την αξία το ότι δεν θα πρέπει να ε, προκαλεί ζημία σε ανθρώπους ή τραυματισμό σε ανθρώπους αλλά ε, στον ποινικό μας κώδικα επιτρέπονται ορισμένες, σε ορισμένες περιπτώσεις σε ανθρώπους να προκαλούν ε, φυσική βλάβη σε άλλον άνθρωπο για παράδειγμα στις περιπτώσεις αυτοάμυνας. Πώς θα εμφυσίσουμε αυτή την αξία σε μηχανή όταν είναι δύσκολο όχι μόνο για τους ε, τεχνικούς αλλά και για μας τους ίδιους να διαλέξουμε αυτές τις αξίες και πώς ακριβώς θα πρέπει να εφαρμόζονται στην πραγματική ζωή. Ε, ευτυχώς βεβαίως συζητάμε για κάτι που ε, θα γίνει στο πολύ απότερο μέλλον αλλά Ίσως θα έπρεπε ως κοινωνία από σήμερα να αρχίσουμε να, να, να εξετάζουμε αυτά τα θέματα. Πρόεδρος, θέλει κάποιος να απαντήσει, κύριε καθηγητά. Πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα και δεν είναι, δεν είναι απλή η απάντηση. Υπάρχουν προβλήματα. Πρώτον πρέπει να προσδιορίσουμε αυτές τις αξίες. Αυτό είναι υποσυζήτηση γιατί μπορεί κανείς να έχει διαφορετικά, ε, ε, διαφορετικές ηθικές προσεγγίσεις σε διαφορετικά προβλήματα. Ίσως θα μπορούσαμε να τα σπάσουμε το θέμα σε συγκεκριμένα ε, επιμέρους προβλήματα τα οποία θα μπορούσαν να συζητηθούν δημόσια στη συνέχεια. Ε, μιλούμε για πλήρως αυτόνομες συσκευές ή μηχανές. Πρέπει κανείς να δει την, αν προσπαθήσει κανείς να λύσει το πρόβλημα συνολικά, ε, θα αποτύχει. Πρέπει να αρχίσουμε σιγά σιγά και κατά περίπτωση να ε, χειριζόμαστε αυτές οι υποθέσεις. Ίσως σε μια πρώτη φάση θα μπορούσαμε ε, σε ένα αρχικό στάδιο να αναθέτουμε σε κάποιον άνθρωπο να επιτηρεί τη λειτουργία μιας συσκευής Υπάρχουν για παράδειγμα τα, οι ηλεκτρικές σκούπες που λαμβάνουν μόνο του αποφάσεις αλλά υπάρχουν και άλλες συσκευές όπου ε, τις μηχανές αυτές που μπορούν με, να λαμβάνουν αποφάσεις τις επιτηρεί, τις εποπτεύει κάποιος άνθρωπος. Αυτό μας υποχρεώνει μέσω κανόνων ή νομικών προτύπων να λύσει πολλά προβλήματα από αυτά που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Φυσικά, το να καταλήξουμε σε πλήρως νοήμονα όντα τα οποία θα μπορούν αυτόνομα να αποφασίζουν και να δρούν, αυτό είναι, είναι, είναι, είναι, είναι πολύ, είμαστε πολύ μακριά ακόμη από αυτό σήμερα. Ε, όταν όμως σήμερα μιλούμε για ε, στρατιωτικά drones, θα ε, μπορούσαν αυτά να λαμβάνουν κάποιες αποφάσεις, αλλά όταν θα έρθει η στιγμή να πατήσει τη σκανδάλη, τότε αυτή την απόφαση να, να πρέπει να την λαμβάνει κάποιος άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε κάποιο κέντρο ελέγχου. Για παράδειγμα, αυτό είναι ένα ζήτημα ε, που το αντιμετωπίζουμε ήδη σήμερα. Η κυρία Κομοντίνη θα μπορούσε να, να δει την ταινία Interstellar μιας και αναφερθήκαμε και στην τέχνη και στα μυθιστορήματα του κυρίου Ασίμου. Ε, η κυρία στο πίσω μέρος της αίθουσας, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η Βάνα Φρούτ από τον Δικηγορικό Σύλλογο της Αγγλίας. Δεν την έχω σκεφτεί ε, διεξοδικά την ερώτησή μου, αλλά ε, θα ήθελα να, να ρωτήσω κάτι σε σχέση με την ευθύνη και την έννοια της αυστηρής ευθύνης που ε, στο πλαίσιο της τεχνητής νοημοσύνης ε, μπορεί να, ε, να επιτελέσει αυτό για το οποίο θεσπίστηκε. Αν όμως υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη που προγραμματιστεί πέραν αυτών των ορίων για παράνομες πράξεις που δεν είχαν προβλεφθεί αρχικώς, τότε ενδέχεται να δημιουργηθούν καταστάσεις αδικίας. Ε, οι ομιλητές έχουν εξετάσει τέτοιες περιπτώσεις. Δεν, δεν ξέρω αν κατάλαβα την ερώτηση. Γιατί όσον αφορά την αυστηρή ευθύνη, σκέφτομαι πάντοτε το ζήτημα της αποζημίωσης. Ε, μιλάμε για αστικές υποθέσεις, όχι ποινικές. Αν όμω η τεχνητή νοημοσύνη προγραμματιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί κανείς να την χρησιμοποιήσει για την διάπραξη ε, παράνομων πράξεων, τότε υπεύθυνο θα είναι εκείνος που προγραμμάτισε τη μηχανή. Γιατί δεν έχει χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο εργαλείο, απλά το χρησιμοποίησε με τρόπο που ε, δεν έπρεπε. γιατί στην ουσία εξαπατώ τους ε, συνανθρώπους μου απλά με ένα πιο προηγμένο τεχνολογικά εργαλείο. Όσον αφορά το ζήτημα της αποζημίωσης, νομίζω ότι το να υπάρχει ένας κανόνας απόλυτης ευθύνης δεν δημιουργεί προβλήματα, διότι θα ξέρει ο, ο εκάστοτε εμπλεκόμενος ότι φέρει την ευθύνη και την, ε, ε, ε, η, ευθύνη για τις επιλογές που κάνει το μηχάνημα θα βαρύνει τον κατασκευαστή ή τον προγραμματιστή. Αυτό εμένα δεν μου φαίνεται ότι θα ήταν άδικο, ακόμη και αν κάποιες φορές θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι η μηχανή θα προβεί σε απρόβλεπτες κινήσεις. Ευχαριστώ. Και επιτρέψτε μου και εγώ να αναφερθώ σε ένα σύνολο κοινών αξιών Θέλω απλώς ε, να σημειώσω ότι πρόκειται για έναν τομέα που χρειάζεται μελέτη. Περαιτέρω, ο Νίκ Μπόστρομ, ο καθηγητής, έχει ιδιαίτερη, ιδιαίτερα μελετήσει τα θέματα αυτά και έχει προσδιορίσει πλαίσια για τις επιλογές και τις συνέπειές τους, αν τα θεωρείτε ενδιαφέροντα νομίζω. Θα βρείτε και απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, μια και δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Θα παρακαλέσω την κυρία Ντελβό να διατυπώσει τα συμπεράσματα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα είναι δύσκολο να διατυπώσω συμπεράσματα. Ευχαριστώ τους ομιλητές μας, τους προσκεκλημένους και το κοινό, όλους αυτούς που έλαβαν μέρος στο σεμινάριο αυτό. Ήταν ε, πολύ πλούσιο σε ενδιαφέροντα, σε έμπνευση. Συζήτησαμε πολλά ζητήματα την αστική ευθύνη, την ασφάλιση, την ηλεκτρονική προσωπικότητα, την κυριότητα των δεδομένων, διαχείριση κινδύνου. Και ρίξαμε και μια ματιά στο μέλλον με την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε αυτή την ομάδα εργασίας για τις νομικές και δεοντολογικές συνέπειες της ρομποτική στην, ομα... στην ε, Επιτροπή μας και συζητούμε τα θέματα αυτά τον τελευταίο χρόνο, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι έχουμε καταλήξει συμπεράσματα, καθώς πολλά νέα προβλήματα ανακύπτουν διαρκώς. Πάντως πιστεύω ότι θα, θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα. Άρα το Μάιο μπορούμε να είμαστε έτοιμοι με την έκθεση. Ε, ήταν πολύ χρήσιμο πάντως αυτά που μας είπατε. Έχουμε να δώσουμε απαντήσεις, έχουμε να κάνουμε ερωτήσεις για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, παραδείγματα drones που κυκλοφορούν ήδη στους εθέρες, τα αυτοκίνητα ε, χωρίς οδηγό, όπου νομίζω θα ήταν σκόπιμο να δώσουμε εμείς ευρωπαϊκές απαντήσεις ε, σε αυτό το πεδίο της εναρμόνισης νομοθεσίας μας σε όλη την Ευρώπη και γι' αυτό πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε περιστασιακά σε πιο άμεσες απαντήσεις και μετά υπάρχουν βέβαια και οι βαθύτερες φιλοσοφικές συζητήσεις και πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο κατάλληλος χώρος να συζητηθούν οι αρχές και οι αξίες που θα πρέπει να καθοδηγούν την έρευνα και την κατασκευή ε, ρομποτικών ε, μηχανημάτων. Μπορούμε και εμείς και οι ερευνητές να διατυπώσουμε προτάσεις. Ο πρώτος στόχος της ε, εκθέσεως θα είναι πρώτα απ' όλα να ευαισθητοποιήσουμε τον πολίτη στο τι είναι μπροστά, τι θα μπορούσε να είναι το μέλλον. Χαίρομαι ιδιαίτερως για την ε, ομάδα εργασίας που έχουμε και την έκθεση. Είναι συναρπαστικό αυτό που έχουμε να κάνουμε. Η συζήτηση συνεχίζεται, δεν κλείνει εδώ. Και σας ευχαριστώ θερμά για την ευκαιρία αυτή τη συζήτηση, προς το παρόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ του ομιλητέ το κοινό, γιατί συμμετείχε στη συζήτηση Θα ξανασυναντηθούμε, είμαι σίγουρος, στο μέλλον.